Good Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ήδη 32 μέλη είναι παρόντα. Θα ψηφίσουμε σήμερα. Και το πρώτο μας σημείο είναι ακριβώς αυτό. Ελπίζω να έχετε όλοι τις κάρτες για την ψηφοφορία μαζί σας. Αρχίζουμε λοιπόν την ψηφοφορία με την πρώτη έκθεση του κυρίου Βάρκαρσελ Σίζο, Πολιτικής Συνοχής και Στρατηγικές Έρευνας και Καινοτομίας για την εφή Εξειδίκευση. Οι στρατηγικές έρευνε και καινοτομία είναι πολύ σημαντικές για την μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής 2013-2020, διότι επικεντρώνονται σε θεματικές και στρατηγικό σχεδιασμό στα πλαίσια του προγράμματος για την ε, εφαρμογή τους επιτόπου. Σε κάθε περιφέρεια θα πρέπει να δούμε τα υπέρ και τα κατά και να δημιουργήσουμε ανάπτυξη βάσει της γνώσης, όχι μόνο σε αναπτυγμένες περιοχές αλλά και σε λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές. Ο κύριος Βαλκαρσέλ ε, παρουσίασε την έκθεσή του. 25 Φεβρουαρίου είχαμε μία προθεσμία για να καταθέσω με 137 κατατέθησαν και ο εισηγητής προτείνει και αρκετές συμβιβαστικές τροπολογίες. Πριν περάσουμε στην ψηφοφορία, θα ήθελε ο εισηγητής να λάβει το λόγο. Κύριε Βάλκαρ Σέλ, θέλετε να λάβετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Θέλω να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας όλους όσους ε, συνεισέφεραν με τις ιδέες τους, με τις τροπολογίες τους κλπ. Πιστεύω ότι το αρχικό κείμενο βελτιώθηκε και εμπλουτίστηκε. Ευχαριστώ λοιπόν όλους όσους βοήθησαν. Ευχαριστώ. Thank you. Thank you very Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στην ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την έκθεση του κυρίου Βαλκαρσέλ και αρχίζουμε με την παράγραφο 1, τροπολογία 26, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 5, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία, τροπολογία 32. Τροπολογία 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή τροπολογία 47 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 48 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 50 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 51 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ κατά αποχές δεκτή 62 υπέρ κατά αποχές δεκτή 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 64 υπέρ κατά αποχές δεκτή 65 υπέρ κατά αποχές δεκτή 66 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 12, συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 71 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 72 υπέρ κατά αποχές δεκτή 73 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή 77 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 14 υπέρ κατά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 96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 97 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 99 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 100 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 101 υπέρ κατά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 αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 114 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 116 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 121. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 122. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 123. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 124. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 19 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 127 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 128 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 129 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 133 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος. Ελέγχουμε την 133. Παρακαλώ. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Είναι δεκτή. Είναι σαφές. Ε, ψηφίζουμε 134 υπέρ κατά αποχές δεκτή 135 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 136 υπέρ κατά αποχές δεκτή 137 υπέρ κατά αποχές δεκτή Τώρα προχωρούμε στις αναφορικές ε, σκέψεις. 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ε, τη σκέψη 11 υπέρ κατά Όχι, είναι η αιτιολογική σκέψη α, η τροπολογία είναι 11 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 12 στην ε, ΑΒ αιτιολογική σκέψη υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 16 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Στην αιτιολογική σκέψη D τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 4. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Στο, στην 25 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, η αιτιολογική σκέψη ΔΕΛΤΑ Και τώρα ψηφίζουμε στο σύνολο της έκθεσης, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε η έκθεση. Συγχαρητήρια κύριε Βαλκαρσέλ. Ωραία. Περνάμε στην έκθεση για την εφαρμογή του θεματικού στόχου ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η έκθεση εφαρμογής για τον συγκεκριμένο στόχο από πλευράς Κομισιόν ε, εστιάζεται στις ε, βασικές προκλήσεις ε, της εφαρμογής του θεματικού στόχου 3 και αναλύει την εφαρμογή της συνέργειας. Αξιολογεί η έκθεση πόσο έχει προχωρήσει η εφαρμογή του συγκεκριμένου θεματικού στόχου, θεματικού στόχου 3, λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες, την αιρεσιμότητα και τη, τα κριτήρια ολοκλήρωσης. Ε, η συγγήτρια η κυρία Ρόζα Νταμάτο υπέβαλε την έκθεση στο Φεβρουάριο, 171 τροπολογίες κατατέθηκαν πριν τη λήξη της προθεσμίας, ενώ η συγγήτρια επίσης προτείνει και στις συμβαστικές τροπολογίες. Θα θέλατε το λόγο. Κύριε Νταμάτο, εδώ δεν είναι, εδώ είναι. Έχετε το λόγο. Θέλω να ευχαριστήσω όσους ε, συνεργάστηκαν μαζί μου, όσες και όσους. Σε αυτή την ε, έκθεση, η οποία μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, ελπίζω ότι ή έχω ικανοποιήσει τους ε, συναδέλφους που υπέβαλαν τροπολογίες. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ κυρία Κρέαλ, έχει θέλει το λόγο. Μια μικρή παράκληση. Υπάρχουν κάποιες τροπολογίες με αριθμούς που δεν είναι σαφής η πηγή. 0,13 μισό τα εκατό ε, σχετικά με τα οχήματα. Εδώ θα πρέπει να γίνει ένας τεχνικός έλεγχος για να δούμε από πού προέρχονται, ποια είναι η πηγή αυτών των αριθμητικών στοιχείων. Αναφέρεστε σε αριθμητικά στοιχεία της έκθεσης ή της, του καταλόγου Όχι, είναι τροπολογίες μου φαίνεται ότι είναι μια από αυτές οι 37 και χρησιμοποιούνται κάποια στοιχεία χωρίς να γνωστοποιείται η, η πηγή. Εγώ δεν μπορώ να τα ελέγξω. Αν ισχύει το περιεχόμενό τους, η ουσία είναι εντάξει. Αλλά θα πρέπει να είναι σωστά τα νούμερα. Οπότε παρακαλώ η γραμματεία να κάνει ένα τεχνικό έλεγχο, ίσως και ο εισηγητής ή η εισηγήτρια μπορούν να κάνουν μια σχετική δήλωση ότι όλα είναι εντάξει. Απλώς δεν θέλω να πάμε στην Ολομέλεια με λάθος νούμερα. Ε, είναι προβληματικό αυτό που ζητάτε, γιατί αν υιοθετήσουμε την έκθεση σήμερα, δεν μπορούμε να την τροποποιήσουμε αργότερα. Αυτός είναι ο κανόνας. Σήμερα ψηφίζουμε την έκθεση. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε το περιεχόμενο. Äh, ναι, αλλά ήθιστε να λέμε στην Ολομέλεια ότι κάποιες τεχνικές προσαρμογές θα πρέπει να γίνουν. Ίσως η κυρία Νταμάτο τώρα μπορεί να κάνει μια σύντομη δήλωση. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρω την προέλευση των αριθμητικών στοιχείων και δεν μπορούσα να το τσεκάρω. Άρα πρέπει να υπάρχει μια δυνατότητα εκ των υστέρων να γίνει ο έλεγχος. Γι' αυτό ήθελα να το ξεκαθαρίσω πριν από την ψηφοφορία, ότι το περιεχόμενο, η ουσία των τροπολογιών είναι απολύτως εντάξει, αλλά ήθελα τα νούμερα να εξεταστούν, να γίνει τεχνική επαλήθευση. Και ε, πριν από την ψηφοφορία και την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα πρέπει αυτό να είναι δυνατόν. Ωραία. Κυρία Νταμάτο, μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο το θέμα αυτό. Σας διαβεβαιώ, συνάδελφε, ότι το προσωπικό, η γραμματεία και όλοι οι συνάδελφοι έχουν τσεκάρει τα νούμερα και βασίζονται σε επίσημες πηγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα, εάν θέλετε περισσότερες διαβεβαιώσεις, και το καταλαβαίνω, θα σας στείλουμε και τα έγγραφα από τα οποία προέρχονται τα δεδομένα, τα αριθμητικά στοιχεία αυτά. Τόσο να έχετε και περισσότερες λεπτομέρειες. Εντάξει, η κυρία Νταμάτο είναι έτοιμη να σας στείλει κυρία Κρέλ τις πληροφορίες αυτές και βέβαια και σε οποιοδήποτε άλλο ενδιαφέρεται με τις συγκεκριμένες αναφορές για τις πηγές των αριθμητικών αυτών στοιχείων. Μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία λοιπόν. Συμβιβαστική πρόταση παριθμών 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική, ε, συγγνώμη, τροπολογία 40 καταπίπτει. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 55. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ. Θέλετε ηλεκτρονική επιβεβαίωση για την 55. Άρχεται η ψηφοφορία για την 55. Λήξη ψηφοφορίας. εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 65. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 67. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η ηλεκτρονική επαλήθευση. Ωραία. Για την 67. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική μόνο μια υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, Συγγνώμη, είχαμε δύο τμήματα, θα επαναλάβουμε την ψηφοφορία. Συμβαστική 9, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική παριθμό 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική παριθμό 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 78 σε δύο τμήματα. Όχι, ε. Ψηφίζουμε μόνο το πρώτο τμήμα υπέρ. Συμβαστική 7. Αφού μου το λέτε, ζητώ συγγνώμη, θα προετοιμαστώ καλύτερα την επόμενη φορά. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Δεν είναι δυνατόν. Ηλεκτρονική επαλήθευση για τη συμβαστική υπαριθμών 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη η ψηφοφορία. Ασφαλώς και υιοθετείτε. Τροπολογία 99. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 101. Δεν θα ψηφίσουμε το πρώτο τμήμα της τροπολογίας 78. Εδώ αναφέρεται ότι αν υιοθετηθεί η, η συμβαστική 6 θα πρέπει να κα, ε, καταπίπτει μόνο το δεύτερο τμήμα της 78, όχι το πρώτο. Σωστά, και εγώ έτσι το είχα διαβάσει, αλλά αλλιώ άλλε οδηγίες μου έδωσαν. Έχετε, συμφω... Έχετε δίκιο. Επιστρέφουμε στην 78. Εδώ έχουμε χωριστή ψηφοφορία, μάλλον ε, κατά τμήματα, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, Ηλεκτρονική επαλήθευση. Πρώτο τμήμα της τροπολογίας 78. Έναρξη ψηφοφορίας. Λήξη. Εγκρίνεται. Οπότε, Προχωράμε στην 101. Σωστά. Ωραία. Τροπολογία 101. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, ε, συμβαστική 20. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική υπαριθμών 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 121 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 13 χωριστή ψηφοφορία πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 134 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 156 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ηλεκτρονική επαλήθευση για την 156 έναρξη ψηφοφορίας. Λήξη. Απορρίπτεται. 157. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 158 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 168 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται.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 αποχές εγκρίνεται. Θεολογική σκέψη Β, τροπολογία 14, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 15, υπέρ, κατά, αποχές. Ε, ηλεκτρονική επαλήθευση. Για την 15. Άρχεται. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική παριθμών 22. Υπέρ. Κατά. Εποχέ. Εγκρίνεται. Συμβαστική 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 25. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση για την 37 έναρξη λήξη ψηφοφορίας εγκρίνεται 38 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τελική ψηφοφορία για το σύνολο του κειμένου. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κυρία Νταμάτου. Τώρα θα συνεχίσουμε με τις δραστηριότητες αντίκτυπο και προστιθέμενη αξία του Ευρωπαϊκού Τομείου προσαρμογής στην προγκοσμιοποίηση μεταξύ 2007 και 2014. Επί της ουσίας είναι η Επιτροπή Απασχόλησης. Κατάρτιση και κινητοποίηση προτείνεται, ο συντάκτης γνωμοδότησης, ακολουθήθηκε γρα... Ε, κατάρτιση γνωμοδότηση και γίνεται μια γνωμοδότηση, έχει γίνει μια μελέτη από ανεξάρτητο σύμβουλο και ε, υπάρχει και η ανακοίνωση της Επιτροπής. Τα δύο έγγραφα στηρίζονται σε δεδομένα από τα κράτη-μέλη για να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος ε, του Ταμείου για την Παγκοσμιοποίηση και να γίνουν και συστάσεις για τη χρήση του. Ο κύριος Ντόιτς είναι ο συντάκτης γνωμοδότησης ε, για τη γνωμοδότηση της Επιτροπής μας τον Ιανουάριο ε, στην συνεδρία της Επιτροπής παρουσιάστηκε 48 τροπολογίες κατατέθηκαν μέχρι την προθεσμία και έγιναν και πέντε συμβιβαστικέ από το συντάκτη της γνωμοδότησης, η ψηφοφορία στην Επιτροπή Απασχόλησης θα γίνει τον Ιούνιο. Προχωρούμε τώρα στην δική μας την ψηφοφορία και αρχίζουμε με τη συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η, η τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 26 Περ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 έχουμε προφορική τροπολογία Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, εξ ονόματος του εισηγητού Τάμας Ντόιτς, θέλω να κάνω την εξής προφορική τεχνικής φύσεως τροπολογία. Θα μπορούσατε να την βρείτε και στο τέλος της ε, αρχική, του αρχικού καταλόγου ψηφοφορίας, αλλά τώρα δεν το βλέπω, οπότε ίσως θα έπρεπε να το διαβάσουμε για να με την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων του Ταμείου και να βοηθήσω με την ταχεία επανενσωμάτωση των άνεργων στην αγορά εργασία, καλεί τα θεσμικά όργανα τη Ένωση, εθνικέ και περιφερειακέ τοπικέ αρχέ να απλουστεύσουν και να επιταχύνουν τη λήψη, τη λήψη αποφάσεων και να εξασφαλίσουν πληρωμέ έγκαιρε από το Ταμείο προ του δικαιούχου επειδή η μέση ε, περίοδος έγκριση είναι 303 μέρες, δηλαδή 10 μήνες και πρέπει να ε, ε, γίνει πολύ μικρότερη κατεπηγόντως για να μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο. Υπογραμμίζει ότι η ενίσχυση των ικανοτήτων των κρατών μελών είναι απαραίτητη ε, ως προς αυτό για να έχουμε καλύτερη συσσόρευση των αποτελεσμάτων και πιο αποτελεσματική. Ωραία. Υπάρχουν αντιρρήσεις? Όχι. Ευχαριστώ. Ψηφίζουμε λοιπόν αυτή την τροπολογία 38 με την προφορική υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Η 39 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Τροπολογία 40 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 41 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 43 υπέρ, κατά, αποχές Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Έλεγχος. Ηλεκτρονικός 43. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Και απερίφθη όντως. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 40. Βεβαίω, 46. Γιατί η 45 έχει αποσυρθεί. Προπολογία 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα τελική ψηφοφορία ε, ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία πέρας η γνωμοδότηση εγκρίθηκε ευχαριστώ πάρα πολύ συνεχίζουμε τώρα με την επόμενη ψηφοφορία η Επιτροπή Μεναφορών συντάσσει μία έκθεση πρωτοβουλίας για, την, για τις μεταφορικές υποδομές στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Εμείς γνωμοδοτούμε απλώς. Μας ενδιαφέρει φυσικά γιατί τα, τα συστήματα μεταφορών είναι σημαντικά για την περιφερειακή ανάπτυξη. Και όσοι ασχολούνται με την περιφερειακή πολιτική θέλουν να βελτιωθούν οι μεταφορικές υποδομές. Ο κύριος Ζέλερ παρουσίασε στις 17 Μαρτίου την γνωμοδότησή του. Έχουμε 51 τροπολογίες και υπάρχουν και συμβαστικές τροπολογίες. Ο κ. Ζέλερ δεν βλέπω να είναι εδώ. Πάμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Ξεκινάμε. Κάτι μου διέφυγε. Κάτι που ήταν αστείο. Ναι, ναι, το πνεύμα του κύριου Ζέλερ είναι εδώ και μας επιβλέπει, ας πούμε. Με την αίσθηση αυτή του πνεύματος του κύριου Ζέλερ ξεκινάμε τη προφορία. Συμβασμός 1, υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. Συμβασμός 2, υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. Τροπολογία 8, υπέρ, κατά Αποχές απορρίπτεται. 9, τροπολογία 9, υπέρ, κατά. Αποχές, υιοθετείται. Τροπολογία 10, υπέρ, κατά. Αποχές, υιοθετείται. Συμβασμός 3, υπέρ, κατά. Αποχές, υιοθετείται. Συμβασμός 4, υπέρ, δύο τμήματα έχουμε εδώ. Ψηφίσουμε το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. Τροπολογία 22, υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. 23, υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. Τροπολογία 26, όχι, ζητώ συγγνώμη, συμβαστική τροπολογία 5, υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. Τροπολογία 32 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Τροπολογία 33 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Συμβασμός 6 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Συμβιβαστική τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές Υιοθετείται. Τροπολογία 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 48 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Τροπολογία 49 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Τροπολογία 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 51 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ψηφίσουμε τώρα το τελικό κείμενο με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετείτε. Μας βοήθησε το πνεύμα του κ. Ζέλερ. Συνεχίζουμε. κυκλοφορούν και άλλα πνεύματα εδώ. Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας, η ΙΤΡΕ, συντάσσει μια έκθεση με βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής με τον ίδιο τίτλο «Έκθεση πρόοδου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας». Κάνει μια ενδιάμεση αξιολόγηση της πρόοδου που έχει γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη προς τους ε, στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας του 2020. Ο κ. Σομερζέμ μας παρουσίασε το σχέδιο νομοθέτησης στην συνεδρίαση του Μαρτίου. Μέχρι την καταληκτική ημερομηνία είχαμε 48 τροπολογίες και ο εισηγητής προτείνει και ε, συμβαστικές τροπολογίες. Ο κύριος Ομερζέ δεν είναι εδώ, δεν μπορεί να παραστεί η σημερινή μας ε, συνεδρίαση. Το πνεύμα του επίσης θα επαγρυπνά. Ξεκινάμε την ψηφοφορία του σχεδίου νομοδότησης. Συμβασμό υπαριθμών 1. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Διαθετείτε. Συμβασμό 2. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Διαθετείτε. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. αποχέ. Πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Την 8. Ψηφίζετε τώρα. Πέρας προφορίας. Υιοθετείτε. Συγγνώμη, τα μπέρδεψα λίγο. Συμβαστική 3 υπέρ κατά. Υιοθετείτε. Τροπολογία 14 υπέρ κατά. Αποχές υιοθετείτε. Τροπολογία 15 υπέρ κατά. Αποχές υιοθετείτε. Τροπολογία 16 υπέρ κατά. Αποχές Απορρίπτεται. Τροπολογία 17. Υπάρχει μια προφορική τροπολογία από τον εισηγητή. Θέλει κάποιος να μας την παρουσιάσει. Όχι. Έχει τις πληροφορίες ούτως ή άλλως για την προφορική αυτή τροπολογία. Υπάρχει κάποιος που είναι κατά. Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν την 17 με αυτή την ε, προφορική τροπολογία. Υπέρ, κατά, αποχές. Υιοθετείται τροπολογία 8, όχι, τροπολογία 18, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε την 18. Την ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. Τροπολογία 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. Συμβαστική τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. Τροπολογία 26. Υπέρ κατά, αποχές, πρέπει να την ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσουμε τώρα την 26 με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Και απορρίπτεται. Τροπολογία 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 28 υπέρ κατά εποχές υιοθετείται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Συμβασμός 6 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Τροπολογία 38 υπέρ κατά αποχές πρέπει να ελέγξουμε φωνικά την 38. Ψηφίζουμε τώρα με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Υιοθετείτε. Τροπολογία 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείτε. Τροπολογία 45 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. Τροπολογία 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και περνάμε στην τελική ψηφοφορία. Ψηφίστε τώρα ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετείτε η γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Πάμε τώρα στη νέα διαδικασία. Εκ μέρους του ΕΛΚ, κυρία Μάλεβιτς ε, έχει μια γραπτή ερώτηση για προφορική απάντηση με συζήτηση σε ό,τι αφορά την επιτάχυνση υλοποίηση πολιτικής συνοχής. Υιοθετήθηκε από τους συντονιστές τον Ιανουάριο και μετά επιβεβαιώθηκε από την Επιτροπή της, ε, από την συνάντηση της Επιτροπής μας. Σύμφωνα με, το, με τις διαδικασίες μας, η κυρία Μάλεβιτς προετοίμασε και ένα προσχέδιο ψηφίσματος, το οποίο μα το παρουσίασε στην περασμένη συνεδρία στο Μάρτιο. Τροπολογίες είχαν προθεσμία μέχρι τι 21 21 Μαρτίου, κατατέθηκαν 47 τροπολογίες. προετοιμάζοντα τη σημερινή ψηφοφορία, οι πολιτικές ομάδες επίση διαπραγματεύτηκαν συμβαστικέ τροπολογίε. Αν υιοθετηθεί το ψήφισμα από την Επιτροπή ή η Γραμματεία, θα το υποβάλει μαζί με το προσχέδιο ερώτησης, το οποίο θα υπογράψει ως πρόεδρος, στην διάσκεψη των πρόεδρων. Η διάσκεψη των Προέδρων θα πάρει την τελική απόφαση για το κατά πόσον η ερώτηση και το σχέδιο ψηφίσματος θα μπουν στην ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας. Κυρία Μάλεβιτς, θέλετε το λόγο. Να σας ευχαριστήσω εσάς και τους συνοδέλφους που στήριξατε το ψήφισμα και για το συμβαστικό πνεύμα όλων. Και ευχαριστώ πολύ που εγκαινιάζουμε έτσι αυτήν την καινούργια διαδικασία. Ωραία. Ξεκινάμε την ψηφοφορία για την προφορική μας ερώτηση και το προσχέδιο ψηφίσματος. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική παριθμών 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασ... Ε, τροπολογία 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική παριθμών 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική υπαριθμών 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική παριθμό 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική υπαριθμόν 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2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 κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το κείμενο στο σύνολό του, άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά, λίγη ψηφοφορία. Ωραία. Εγκρίναμε αυτή την προφορική ερώτηση και το σχέδιο ψηφίσματος και τελειώνουμε τις ψηφοφορίες έγκαιρα. Ευχαριστώ πολύ για τη στήριξή σας. Συνεχίζουμε το επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης. Our next item of business. Ε, το σχέδιο για την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή των Άλπων. Η στρατηγική αφορά 7 χώρες, 5 εκ των οποίων είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι κράτη-μέλη. Και δύο δεν είναι κράτη-μέλη οκτώ περιφέρειες περιλαμβάνονται σε αυτή τη στρατηγική και η συνολική κατοική της περιοχής των Άλπαιων είναι πάνω από 18 εκατομμύρια. Καλύπτονται τρεις θεματικές ε, πολιτικές, ε, κινητικότητα, περιβάλλον, οικονομία. Η, ε, η έκθεση πρωτοβουλίας εστιάζει το δυναμικό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες δυνατότητες χρηματοδότησης με στρατηγικό σχεδιασμό και αστικών και εξωστικών περιοχών. Επίσης, απαιτεί από τα κράτη-μέλη, ζητεί από τα κράτη-μέλη. Μπορώ παρακαλώ πολύ να σας ζητήσω να κάνετε λίγο περισσότερη ησυχία φεύγοντας. Ωραία. Η, η μα είναι η κυρία Μπρέσο. θα μας παρουσιάσει το προσχέδιο εκθεσή της. Η ε, προθεσμοί για τις τροπολογίες είναι στις 5 το απόγευμα την 3η 26 Απριλίου. Θα σας το υπενθυμίσω κιόλας. Δίνω το λόγο στην κυρία Μπρέσο. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να σας υπενθυμίσω ότι σας διέφυγε ή μας διέφυγε να προσθέσουμε στην πρώτη παράγραφο της έκθεσης ότι μιλάμε για τις γενικές παρατηρήσεις, ότι υπάρχει και το θέμα της ε, διακυβέρνησης ή διαχείρισης, του governance, γιατί είναι ένα από τα τέσσερα σημεία της στρατηγικής. Θα το βάλουμε όμως, θα το εντάξουμε χάρη στις τροπολογίες. Λοιπόν, η έκθεση, όπως υπενθυμίσατε, αφορά την πρώτη μακροπεριφερειακή στρατηγική που δεν αφορά ποτάμια ή θάλασσες, αφορά μια μεγάλη ορεινή περιοχή των Άλπαιων. Δεν αφορά όμως μόνο τον ορεινό όγκο αυτό καθεαυτό, αλλά και τις περιαλπικές περιοχές, καθώς και τις πεδιάδες γύρω-γύρω. Επομένως, μιλάμε για μια τεράστια πρόκληση, για ένα στρατηγικό project που ενώνει για πρώτη φορά τις ορεινές περιοχές των Άλπαιων με τις άλλες που είναι πολύ αναπτυγμένες και που περιτριγυρίζουν τις Άλπεις. Μεταξύ των οποίων υπήρχε πάντα ένας μεγάλος διάλογος. Λόγω του ότι είναι τεράστιος αυτός ο χώρος, 80 ε, εκατομμύρια άνθρωποι, 48 περιφέρειες κτλ, 7 κράτη, το θέμα της governance είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως σημαντικό είναι και ότι τα διαρθωτικά ταμεία και τα επενδυτικά ταμεία που εγκρίθηκαν πριν από την έγκριση της στρατηγικής θα πρέπει να συγκλίνουν κατά τη χρησιμοποίησή τους προς ε, κοινά εργαλεία για την ανάπτυξη αυτής της περιοχής. Είναι σημαντικό και τα διάφορα όμως ευρωπαϊκά ταμεία, τα οποία δεν αφορούν την στρατηγική των Άλπιων, αλλά που θα μπορούσαν να προσανατολιστούν και μέσω ειδικών προγραμμάτων για να αφορούν και την ε, περιοχή των Άλπαιων, να λάβουν υπόψη λοιπόν την στρατηγική, το COSME, το Horizon κτλ. Η έκθεση λέει ότι η Κομισιόν θα πρέπει να εξετάσει την προστιθέμενη αξία των, ε, και τις προκλήσεις που αφορούν την περιοχή αυτή. Ένα άλλο σημαντικό σημείο αυτών των γενικών παρατηρήσεων που αφορά τον governance είναι ότι ζητούμε από το Κοινοβούλιο να εμπλακεί ε, στο USALP που είναι το διαχειριστικό όργανο και η Κομισιόν να παίξει ένα εργό ρόλο. Όχι μόνο να συντονίζει και να υποστηρίζει ας πούμε το USALP και να εγκριθεί η εφαρμογή ε, με δείκτες ε, μετρήσιμους και για το θέμα της governance και κάτι άλλο να πω. Μια και οι πρωτεύουσε των κρατών των Άλπαιων είναι πολύ μακριά από την καρδιά της αλπικής περιοχής, στη φάση της ενεργοποίησης, το governance να είναι περισσότερο στα χέρια των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Και στις πολυάριθμες ομάδες των ενδιαφερομένων, των stakeholders που ασχολούνται για να αναπτυχθεί η περιοχή. Με την αρχή λοιπόν με σεβασμό της, αρχική, της αρχής της επικουρικότητας και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Η στρατηγική διαρθρώνεται γύρω από τρεις μεγάλους θεματικούς άξονες. Η οικονομική ανάπτυξη και η καινοτομία είναι ο πρώτος άξονας και καλούμε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μαζί με την Κομισιόν να αξιολογήσει τη δυνατότητα να δημιουργήσει μια συγκεκριμένη πλατφόρμα επενδύσεων ad hoc, ειδικά για τις Άλπεις, αξιοποιώντας και τα ταμεία της Ευρωπαϊκής ε, Τράπεζας Επενδύσεων, αλλά και τα κονδύλια που υπάρχουν από το σχέδιο Juncker, ούτως ώστε να δημιουργηθούν διάφορα project που θα χρησιμοποιούν αυτή την πλατφόρμα για να προσελκύσουν επενδυτές. Δεύτερον, Υπάρχουν διάφορα θέματα. Δεν έχω χρόνο τώρα να τα αναφέρω λεπτομερώς, αλλά ξεκινούν από την αρχή ότι η περιοχή των Άλπαιων δεν είναι μόνο μια περιοχή όπου οι παραδόσεις ε, πρέπει να διατηρηθούν. Οι παραδοσιακέ δραστηριότητε ε, θα πρέπει να αξιοποιηθούν και να διατηρηθούν, αλλά είναι και μια τεράστια περιοχή και ένα φυτόριο, α πούμε, Αυτή η μακροπεριφέρεια των Άλπαιων έχει πάρα πολλά πανεπιστήμια, πάρα πολλά ερευνητικά κέντρα η καινοτομία, οι νέες τεχνολογίες δεν λείπουν και από αυτή την ε, περιφέρεια που είναι ε, παραγωγός ε, καινοτόμων ιδεών. Ενθαρρύνουμε λοιπόν τη συνεργασία, ούτω ώστε να δημιουργεί ένα πραγματικό δίκτυο με αυτέ τι δραστηριότητε, γύρω από αυτέ τι δραστηριότητε, με, με κέντρο τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα, αλλά και διάφορε επιχειρήσει και διάφορου ενδιαφερόμενου, ούτω ώστε να γίνει πραγματικό πόλο καινοτομία η περιοχή. Μιλάω κυρίω για τεχνολογίε καινοτόμε και βιώσιμε, λαμβάνοντα υπόψη τη σημασία του περιβάλλοντο, ειδικά σε αυτή την ε, στρατηγική. Σε ό,τι αφορά τις τουριστικές δραστηριότητες κυρίως, αλλά και όλες τις παραδοσιακές δραστηριότητες των ορεινών περιοχών, η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα και τονίζω, τα τονίζω πάρα πολύ στην εκθεσή μου. Στη δεύτερη παράγραφο, ή μάλλον το δεύτερο θέμα της στρατηγικής, αφορά την κινητικότητα και την διασύνδεση. Εδώ οπωσδήποτε πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι τα συστήματα μεταφορών στις περιοχές των Άλπιων και τις περιαλπικές περιοχές, λόγω της γεωγραφίας των εδαφών αυτών, είναι πάρα πολύ δύσκολο θέμα, πάρα πολύ περίπλοκο. Και σε πολλές περιφέρειες το σύστημα μεταφορών, το τοπικό, είναι εντελώς ανεπαρκές. Γιατί είναι περιοχές που τις διατρέχουν μεγάλοι ευρωπαϊκοί άξονες, τα μεγάλα TNT, τα μεγάλα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών δηλαδή. Όμω η διασύνδεση μεταξύ αυτών των μεγάλων αξώνων και το εσωτερικό σύστημα μεταφορών στις ε, υποπεριοχέ είναι πάρα πολύ σημαντικό, ούτω ώστε να μπορούν να αξιοποιούνται όλες οι ευκαιρίες που υπάρχουν από τη διασύνδεση. Και καινοτόμε ε, μορφές μεταφορών που χρησιμοποιούν επίσης και το sharing economy θα μπορούσαν να είναι χρήσιμο σε περιοχέ όπου οι παραδοσιακές δημόσιες μεταφορές δεν αντέχουν, δεν είναι αρκετές. Παρότι βεβαίως, εκεί όπου έχει, δεν παίζει το ρόλο της η αγορά, ε, δεν υπάρχουν αρκετές επενδύσεις κτλ. Δεύτερο πρόβλημα είναι οι δυσκολίες και η ανεπαρκής ψηφιακέ διασυνδέσει σε πολλέ περιοχέ. Αν θέλουμε πραγματικά να γίνει πολλή χιονοτομία η περιοχή και να γίνει πολύ εξυγχρονισμένη περιοχή, προφανώ θα πρέπει οι δημόσιε αρχέ να παρεύουν και να βελτιώσουν την ε, διασύνδεση με επενδύσει που είναι δυνατέ, γιατί μερικές φορές σε αυτές τις ζώνες η αγορά τα έχει φτύσει ούτως ε, επομένως, οι δημόσιες ε, επενδύσεις ε, στις ορεινές περιοχές είναι ένα άλλο σημείο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και το αναφέρει πολύ συγκεκριμένα η έκθεση. Το τρίτο στατηγικό θέμα, το οποίο επιλέγει από την USALP, είναι το θέμα της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Είναι μια τεράστια κληρονομιά βιοπικιλότητας η Άλπης. Πρέπει να την προστατεύσουμε, αλλά και να βάλουμε και να εισαγάγουμε και καινοτόμα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, κυρίως την προστασία που συνδέεται με τη στρατηγική για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρήπανσης, όπου στις περιοχές της παιδινές είναι ιδιαίτερα έντονο λόγω των χαρακτηριστικών του κλίματος. Δεν, υπάρχουν, ε, δεν υπάρχει αρκετός αέρας, ας πούμε, στα στους πρόποδες των, του βουνού ας πούμε και υπάρχει πρόβλημα λοιπόν, υπάρχει μόλυνση. Ε, θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την α, ατμοσφαιρική ρήπανση ώστε να προστατεύσουμε και τη βιοπικιλότητα. Επίσης υπάρχουν διάφορα ορεινά πάρκα και παιδινά πάρκα και θα πρέπει να δουλέψουμε ούτως ώστε να προστατεύσουμε την βιοπικιλότητα και να υπάρξει και μια διασύνδεση ανάμεσα στις διάφορες προστατευόμενες περιοχές. Φυσικά είναι μια περιοχή που προσφέρεται για την ε, αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από, ε, από την υδροηλεκτρική ενέργεια που είναι πιο παραδοσιακή, αλλά έχει ακόμα περισσότερο δυναμικό, ε, αιωλική ενέργεια, η, ε, ηλιακή ενέργεια, χρησιμοποιώντας και τις, το δυναμικό των δασών επίσης. Πρέπει να τονίσουμε τη σημασία της δουλειάς που έχει κάνει η υπηρεσία παρακολούθησης ε, του Χάλιβα μετά ε, από, τις, από το COP21 και από τις στρατηγικές που αποφασίστηκαν. Συγγνώμη, η Επιτροπή Παρακολούθησης συγγνώμη, των παγετώνων. Των παγετώνων, όχι του Χάλιβα. Και υπάρχει πρόβλημα γιατί ε, είναι σημαντικό να μειωθεί το διοξείδιο του άνθρακα γιατί ε, μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ τους παγετώνες. Όλες οι χώρες, οι περιφέρειες και οι τοπικές αρχές θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή την ε, διαφοροποίηση ενεργειακού ανεφοδιασμού και ούτω ή άλλω η αλλω η ενέργεια εκεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο υπόλοιπο των χωρών αυτών, των 7 αυτών χωρών τη περιοχή των Άλπαιων. Νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά σημεία. Δεν είχα πάρα πολύ χρόνο, Ούτω ή άλλω ε, ξεπέρασε τον χρόνο που μου δόθηκε. Θέλω να υπενθυμίσω σε όλου του συναδέλφου ότι θα κάνουμε την Πέμπτη το πρωί μία συνάντηση με τους σκιώδει εισηγητέ, ούτω ώστε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση τη νομοδότησης εν γέννη και να δούμε αν υπάρχουν στοιχεία τα οποία λείπουν κατά από των σκιωδών εισηγητών και τα οποία θα πρέπει να εντάξουμε στην έκθεση. Και με, βάλει, και με βάση τις τροπολογίες θα βάλω και στην έκθεση λαμβανωμένων υπόψη των ορίων που έχουμε, γιατί δεν, δεν έχουμε απεριόριστο χώρο στην έκθεση, θα βάλω διάφορα άλλα στοιχεία που θα τα θέλουν οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Αρχίζουμε τη συζήτηση τώρα. Πρώτα οι σκιώδες. Για το ΕΛΚ, κυρία Σμιτ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και την εισηγήτρια για μια έκθεση που όχι μόνο εγώ αλλά και οι συνάδελφοι της ομάδας μου θεωρούν πολύ καλή, λεπτομερή διεξοδική, από την αρχή θα έπρεπε να μην δοθούν περισσότερα χρήματα, ούτε να δημιουργηθούν περαιτέρω επίπεδα διοίκησης. Αυτό δεν συμβαίνει. Είπατε ότι το θέμα αφορά 7 ε, χώρες, 48 περιφέρειες, 80 εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτοί είναι άνθρωποι που ασχολούνται και με άλλα θέματα του αλπικού χώρου, εντατικά στις περιφέρειές τους και στις χώρες τους και ήρθε πια η ώρα και νομίζω ότι η έκθεση αυτή είναι καλή ευκαιρία ήρθε πια η ώρα να ανταμυφθούν σε εισαγωγικά οι άνθρωποι αυτοί και πώς θα γίνει αυτό, στηρίζοντας τα project, τα έργα που έχουν προχωρήσει. Όχι με έργα μόνο, αλλά με... όχι μόνο με λόγια, αλλά με έργα. Βέβαια, χρειάζονται και κάποιες ε, οικονομικές ε, ε, πρικοδοτήσεις. Από τη μία πλευρά, όπως είπε η συγγήτρια, μέσω της πλατφόρμας αυτής, ε, μέσω της ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, αλλά και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναγνωρίσουν ότι τα επενδυόμενα στον αλπικό χώρο χρήματα θα ωφελήσουν ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα διευρωπαϊκά διοίκτυα στον τομέα των μεταφορών κυρίως περνούν από τις Άλπεις. Αλλιώς δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. Όλοι προφανώς θέλουμε έναν αλπικό χώρο πολύ με βιοπικιλότητα που θα προστατεύει τη φύση, αλλά και από την άλλη πλευρά δεν θέλουμε να εξακολουθούν να ε, εξαναγκάζονται οι νέοι να φεύγουν από τις μεγάλες πόλεις. Θέλουμε να βρεθεί δυνατότητα να παραμείνουν στις κοιλάδες των Άλπαιων και στις παιδινές περιοχές να βρουν επαγγελματική δραστηριότητα και μέλλον εκεί. Οπότε θα πρέπει να υπάρχουν διασυνδέσεις στις μεταφορές, αλλά και με βριζονικές διασυνδέσεις κλπ. Και σε άλλους τομείς να υπάρχει διασύνδεση, να εξασφαλιστεί αυτή. Αλλιώς δεν θα τα καταφέρομαι και στο μέλλον θα έχουμε παιδιάδες και κοιλάδες των Άλπαιων ε, ερημωμένες, χωρίς πληθυσμό. Ξέρουμε ότι πολλές περιοχές που ζουν αποκλειστικά από τον τουρισμό δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν αυτή τη δραστηριότητα και στο μέλλον. Ο τουρισμός είναι σημαντικός, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και στις ε, διασυνδέσεις των μεταφορών, αλλά δεν μπορούμε νομίζω στο μέλλον αποκλειστικά να βασιζόμαστε στον τουρισμό, αλλά να δημιουργήσουμε κίνητρα και για άλλα επαγγέλματα να ανθίσει η οικονομία και σε άλλους τομείς στον χώρο των Άλπαιων και να παραμείνει η οικονομία εκεί, ούτως ώστε να εξασφαλιστούν θέσεις εργασίας για τους διαμένοντες εκεί και να έχουν οι τελευταίοι κίνητρα να παραμείνουν σε αυτές τις περιοχές. Είναι πολύ σημαντικό στην έκθεση και το έχω ζήσει και εγώ γιατί και στη χώρα μου εγώ είμαι Αυστριακή και έχω συζητήσει και με πολιτικούς ε, στο περιφερειακό επίπεδο, ε, διοικητικά στελέχη κλπ. Και μου λένε ότι είναι σημαντικό η δουλειά να γίνει από κάτω προς τα πάνω, να μην ε, υπαγορευτούν οι λύσεις άνωθεν, αλλά στις περιφέρειες ο κόσμος που ζει να ξέρει και να καταλαβαίνει και να παρακολουθεί. Και να συμφωνεί βέβαια για, σχετικά με το τι θα γίνει στο χώρο του, στο χώρο των Άλπαιων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και έχει δίκιο η εισηγήτρια που λέει ότι πρέπει να ε, συμμετέχει και το Κοινοβούλιο, όχι μόνο εγκρίνοντας την έκθεση, που αυτό έτσι όπως ε, θα γίνει δεν θα συνεπάγεται μεγάλο αντίκτυπο, αλλά θα πρέπει να ε, δράσουμε αποτελεσματικά, να λάβουμε υπόψη μας όχι μόνο τις κοιλάδες αλλά άλλες περιοχές και να ενισχύσουμε μαζικά τη διασύνδεση των Άλπαιων και να εξασφαλίσουμε ότι ο χώρος των Άλπαιων όχι μόνο για τις ε, συγκεκριμένες χώρες αλλά για όλη την Ευρώπη θα έχει μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λούερ είναι ο επόμενος ε, ε σκιώδης. Α, α, α, με συγχωρείτε. Ο, ο κύριος Σερνατζότο. Έχετε το λόγο. Δύσκολο επώνυμο έχω, το ξέρω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την πολύ καλή της έκθεση, η οποία λαμβάνει υπόψη κυρίως την ανάγκη ανάπτυξης αυτής της περιοχής. Εγώ μιλάω την καθεαυτό αλπική περιοχή, όπου τα τελευταία 10-15 χρόνια έφυγε πολλοί κόσμος και υπάρχει, υπάρχουν περιοχές που εγκαταλείφθηκαν, ε, γιατί έχουμε μόνο παθητικές υποδομές στην περιοχή. Είναι μία από τις δύο πιο σημαντικές ε, παραγωγικές περιοχές της, της, της Ευρώπης. Ε, την κοιλάδα του, μαζί με την κοιλάδα του Πάδου και την κοιλάδα της Βαβαρίας. Θα πρέπει να σταματήσουν αυτές οι παθητικές υποδομές και να υλοποιηθούν ενεργητικές υποδομές. Τι σημαίνει αυτό, ότι αν υπάρχει μία μεταφορά προς, ε, και υπάρχει ένας διάδρομος ε, η ο παραγόμενος πλούτος επενδύεται εκεί, ας πούμε, για την προστασία του περιβάλλοντος, για όλο τον πλούτο που ξέρουμε, ας πούμε. Και έτσι σταματάει αυτή η ανάπτυξη παθητικών υποδομών. Γι' αυτό διαβάζω με μεγάλη ικανοποίηση διάφορα σημεία της έκθεσης Μπρέσο. Θα υποβάλω και κάποιες μικροτροπολογίες, αλλά τίποτα σημαντικό, γιατί ουσιαστικά τα έχει όλα. Μιλάει για την ανάπτυξη της κεντρικής περιοχής που παράγει ευημερία και ποιότητα ζωής. Και αυτό θα πρέπει να μεταφερθεί και να υπάρχει μια διασύνδεση με αυτές τις περιοχές και τις ε, παιδιάδες. Εγώ ζω στην κοιλάδα του Πάδου, που είναι η πιο μολυσμένη της Ευρώπης ίσο. Στα νότια των Άλπαιων. Η φύση από μόνη της δεν μπορεί όλα αυτά που παράγονται ε, σε μια περιοχή που είναι πολύ παραγωγική, που έχει πάρα πολύ κόσμο κτλ. Δεν μπορεί να καθαρίσει η φύση από μόνη τη, πούμε, το περιβάλλον. Και νομίζω ότι αυτά τα λέει η έκθεση. Ο, ο διάδρομος ε, όταν είναι μόνο άσφαλτος απλώς, ε, ένα διάδρομος από άσφαλτο μπορεί να φέρει και μία κάποια έτσι αμηχανία αλλά σίγουρα και ευημερία. Είναι λοιπόν μια τεράστια ευκαιρία, όχι μόνο για την ανάπτυξη και την διατήρηση και την ανάπτυξη του πληθυσμού στην περιοχή των Άλπων, αλλά για την ευημερία και την ποιότητα ζωής ε, και στο, στις Βόρειες Άλπες αλλά και στις Νότιες Άλπες. Ευχαριστώ. Ο κ. Γιάκοφτσιτς, επόμενος και ο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους και όλους Θέλω καταρχήν να συγχαρώ την κυρία Μπρέσο. Η έκθεση της είναι Και χαίρομαι που συμμετέχω και εγώ στην επεξεργασία της. Ως εισηγητής ε, για την ε, στρατηγική για την Αδριατική και το Ιόνιο, θέλω να υπογραμμίσω το εξής είχαμε αποφασίσει να χρησιμοποιήσουμε την ε, προσέγγιση των τριών όχι. Αυτό θα πρέπει να συζητηθεί πολύ σοβαρά. Στη στρατηγική για το Ιόνιο και την Αδριατική. Αν δεν διαθέτουμε μια ελάχιστη συντονιστική δομή, δύο-τριών ατόμων, δεν λέω τίποτα παραπάνω, στις Βρυξέλλες ή κάπου αλλού, στην ίδια την μακροπεριφέρεια, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Χρειαζο... Έχουμε πόρους. Αυτό που λείπει όμως είναι ο συντονισμός των διαφόρων έργων και προγραμμάτων που είναι διαθέσιμα για τη χρηματοδότηση. Κάποιος θα πρέπει να συνεχίσει το έργο που ξεκινήσαμε. Και μία από τις αδυναμίες των μακροπεριφερειακών στρατηγικών γενικότερα είναι αυτή. Όπως είπε και ο πρώμος ομιλητής, υπάρχει θέμα επικοινωνίας εντός της αλπικής περιφέρειας μεταξύ του βορρά και του νότου και προς την περιφέρεια αυτή. Εγώ συχνά οδηγώ από την Κροατία στο Στρασβούργο και περνώ από την αλπική περιφέρεια. Και μπορώ να σας πω από προσωπική εμπειρία ότι πολλά απομένουν να γίνουν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πλήρως το δυναμικό της ε, περιφέρειας αυτής. Στηρίζω την έκθεση και πιστεύω ότι ε, πολλά από αυτά που αναφέρει είναι πολύ σωστά. Για παράδειγμα, ε, τα σχετικά με την οικονομική ανάπτυξη, αλλά και άλλα. Θα πρέπει να δούμε πώς θα βασιστούμε σε αυτή τη στρατηγική, να χτίσουμε και ιδιαίτερα στο θέμα της επικοινωνίας μεταξύ του βόρειου και του νότιου τμήματος της αλπικής περιφής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω κυρία Μπρέσο Είναι πολύ σημαντικό ε, σίγουρα να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματική διακυβέρνηση της περιφέρειας. Όπως είπε ο κ. Γιάκοψιτς, ε, είναι πολύ σημαντικό ε, και οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να υλοποιούνται με βιώσιμο τρόπο. Τα κράτη-μέλη που ανήκουν σε αυτή την περιφέρεια θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα κονδύλια Είτε πρόκειται για ευρωπαϊκά κονδύλια, είτε πρόκειται για ιδιωτικά. Επιπλέον, χαίρομαι που η συγγήτρια αναφέρει κάποια πολύ σημαντικά πράγματα, όπως η προστασία της βιοπικιλότητας, η σημασία της, ε, της συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την καινοτομία. Και ως αισιόδης ηγητής για την κυκλική οικονομία από πλευράς Επιτροπής Περιβάλλοντος, Θέλω να υπογραμμίσω τη σημασία της κυκλικής οικονομίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να αλλάξουμε την προσέγγιση μας σε ό,τι αφορά την κυκλική οικονομία. Πρέπει να προστατεύσουμε τις τοπικές και περιφερειακές οικονομίες. Θα πρέπει να συμπεριλάβουμε την κλιματική αλλαγή σε όλα τα επιχειρηματικά μας μοντέλα. και να χρησιμοποιούμε τους φυσικούς ε, πόρους πολύ προσεκτικά και με σύνεση. Ε, και προφανώς να ευαισθητοποιήσουμε και το κοινό γι' αυτό. Ο δημόσιος τομέας ε, πρέπει να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας, ιδιαίτερα μέσω των κρατικών προμηθειών, έτσι ώστε να, προστατέ να προωθήσει την κυκλική οικονομία και την πράσινη οικονομία γενικότερα. το παραγωγή ενέργειας επίσης σε τοπικό επίπεδο είναι σημαντική όχι μόνο γενικότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ειδικότερα για την αλπική ζώνη. Χρειαζόμαστε τεχνολογία και προγράμματα, σχέδια μάλλον, έργα, τα οποία θα είναι προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες. Η ενεργειακή, ο ενεργειακός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ενεργειακή επάρκεια και θα πρέπει να δώσουμε βάρος στην τοπική παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Αυτό συνδυάζεται και με την καταπολέμηση της φτώχειας. Η αλπική περιφέρεια είναι η δεύτερη μεγαλύτερη περιοχή βιοπικιλότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τεράστια, ε, τεράστιες εκτάσεις οι οποίες θα πρέπει να προστατευτούν μαζί με τα οικοσυστήματά τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για τις ιδέες που έχει βάλει στην έκθεση. Συμφωνώ με τις προηγούμενες ε, παρεμβάσεις. Όλοι συμφωνούμε ότι η αλπική περιοχή είναι μια κληρονομιά βιοπικιλότητας που πρέπει να διατηρηθεί τα επόμενα χρόνια, δεκαετίες κτλ. Αυτό είναι το σημείο αφετηρίας για να δούμε τι δράση θα πρέπει να προωθήσουμε. αυτή η περιοχή θα πρέπει να θεωρηθεί ως εργαστήρι ανάπτυξη για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκινώντας από αυτή την έκθεση μπορούμε να αλλάξουμε λιγάκι την προσέγγιση που έχουμε για την ε, περιοχή αυτή. Μία προσέγγιση ε, η οποία θα πρέπει να στοχεύει στην αξιοποίηση των καλών πρακτικών ε, για την προστασία του, των φυσικών αγαθών, το, του νερού, του εδάφους, τη διατήρηση του εδάφους, και να έχουμε και νέα συστήματα ε, μέτρησης της πρόοδου. Όχι μόνο να βασιζόμαστε σε οικονομικούς δείκτες, αλλά και σε κοινωνικούς δείκτες. Προσοχή στις δράσεις που θα αναπτύξουμε. Θα πρέπει να δούμε τι πραγματική επίπτωση έχουν οι δράσεις αυτές στο περιβάλλον. Όχι απλώς να προστατεύουμε το περιβάλλον, αλλά και όλο το κοινωνικό-οικονομικό σύστημα από το οποίο εν συνεχεία εξαρτάται ολόκληρη περιοχή. Και επίσης οι αποφάσεις δεν πρέπει να έρθουν άνωθεν. Θα πρέπει να έχουμε διάφορους μηχανισμούς άμεσης διαβούλευσης, το είπαμε πάρα πολλές φορές, να έχουμε στρατηγικές που ξεκινάνε από κάτω και πηγαίνουν προς τα πάνω. Στο κέντρο λοιπόν αυτής της δράσης εμείς θα πρέπει να εντάξουμε ε, έννοιες όπως η βιωσιμότητα και ο προγραμματισμός, ο σχεδιασμός. Αυτό είπαμε όλοι μας όσοι πήραμε το λόγο για αυτή την έκθεση. Θα ήθελα να κάνω και κάποιες παρατηρήσεις όμως για τα επώδυνα σημεία. Τι γίνεται δηλαδή όταν περνάμε από τα λόγια στα έργα. Συχνά μιλάμε για τη χρήση των Ευρωπαϊκών Ταμείων. Είναι εκ των όνου αυτά τα ταμεία αυτά και είναι πολύ καλά γιατί και η οικονομική διάσταση είναι πάρα πολύ σημαντική για να μπορέσει να επανεκκινήσει η οικονομία μιας περιοχής. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να καταλάβουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα κονδύλια, αλλά προς ποιου στόχους. Γιατί η αίσθησή μου είναι ότι πέρα από τα λόγια τα οποία γράφει η έκθεση, δημιουργούμε μετά ιδέες, ούτως ώστε η προσοχή μετά να πάει στα μεγάλα έργα. Που όμως είπαμε ότι συχνά είναι έργα τα οποία έχουν σαν σκοπό να δημιουργήσουν άξονες ας πούμε για να περάσει ο κόσμος από εκεί αλλά όχι για να παραχθεί πλούτος ας πούμε που θα μείνει και στην περιοχή. Μιλάμε για γραμμές υψηλής ταχύτητας, για μεγάλους άξονες οδικούς κτλ. Πριν χρηματοδοτήσουμε νέα έργα, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τα υπάρχοντα και να τα καταστήσουμε αποτελεσματικά. Συχνά τα υποχρησιμοποιούμε. Αν μιλάμε για ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, ούτω ώστε ε, να μην δοθούν κίνητρα για να προωθηθούν δράσεις, ας πούμε, κερδοσκοπίας. Μιλάω για πρακτικές που έχουμε δει σήμερα στον τομέα της υδροηλεκτρικής ενέργειας. Δημιουργείται πλούτος ο οποίος φεύγει στο εξωτερικό και δεν ε, μένει ούτε στην περιοχή αυτή, ούτε επωφελείται ο τοπικός πληθυσμό. Τέλος, για την διάσταση της περιοχής, της περιφέρειας, μία παρατήρηση. Η περιοχή των Άλπων, έτσι όπως την εντοπίσατε, είναι μία τεράστια εκθεση Μιλάμε για 80 εκατομμύρια κατοίκους που μένουν εκεί. Αυτό μπορεί να είναι και ενδιαφέρον από μία πλευρά έτσι, και συγκλονιστικό, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε. Μία τόσο αχανής περιοχή καλύπτει υποπεριφέρειες με διαφορετικά προβλήματα. Και συχνά ε, οι, περιο... οι αυτές δεν γίνονται με την ίδια ταχύτητα. Δεν θα θέλαμε λοιπόν με την ε, δικαιολογία ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε βάσεις για δράσεις οι οποίες ε, αφορούν όλη την περιοχή. Τελικά οι συγκεκριμένες δράσεις να δημιουργήσουν προβλήματα και να ζημιώσουν τις υποπεριοχές που έχουν τελείως διαφορετικές ανάγκες. Ευχαριστώ. Η κυρία Κρέλλη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Η έκθεση, το σχέδιο έκθεσης μας ε, υπέβαλε είναι πολύ καλό. Άπλεται πολλών τομέων που ε, είναι σημαντική, μπορεί να αποκούν σημαντική στην περιοχή των Άλπαιων. Το σχέδιο είναι πολύ καλό. Εγώ ζήτησα το λόγο για να αναφέρω το θέμα της πρόσθετης χρηματοδότησης. Τα κονδύλια που έχουμε στη διάθεσή μας για την πολιτική συνοχή στα κράτη-μέλη για τέτοιες ε, μακροπεριφερειακές στρατηγικές πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε περισσότερο και μπορούμε να συνεργαστούμε και διασυνοριακά και να τα δώσουμε και για την περιοχή των Άλπαιων. Πρέπει όμως να προσελκύσουμε και ιδιωτικά κεφάλαια, ούτω ώστε το αποτέλεσμα να ξεπερνά το τι μπορεί να προσφέρει η πολιτική συνοχή. Μια μικρή προειδοποίηση, αν και δεν είμαι σίγουρη αν η σκιώδηση συγκεκριμένα εννοούσε έτσι σε σχέση με τα νέα κονδύλια από τα ευρωπαϊκά ταμεία για τι μακροπεριφερειακές στρατηγικέ για τη διάθεση αυτών των κονδυλίων. Εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος. Δηλαδή, να ε, βάλουμε ο ένας τρικλοποδιά στον άλλον. Εμείς ε, στο δημοσιονομικό πλαίσιο δίνουμε καθημερινά μάχη για μια σωστή πολιτική συνοχή. Είναι το 1 τρίτο του ενωσιακού προϋπολογισμού και πολλοί και ευρωβουλευτές θα ήθελαν τα χρήματα αυτά να δοθούν σε άλλα έργα. Αν στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής πούμε ότι θέλουμε περισσότερα κονδύλια για τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές θα δημιουργηθεί κατάσταση ανταγωνισμού. Γιατί ξέρω ότι ποιοι είναι αυτοί που περιμένουν ε, να κάνουν στρατηγική και σε άλλους τομείς. Ε, υπάρχουν και άλλα πάρκα, υπάρχουν και άλλα ποτάμια, υπάρχουν ε, και άλλες περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν να, μείνουμε να παραμείνουμε αυστηροί. Η συνεργασία μεταξύ κρατών μελών θα πρέπει να προωθηθεί και συνεργασία με τρίτες χώρες, ούτω ώστε οι πόροι που υπάρχουν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικότερα πάνω στη βάση μιας κοινής στρατηγικής για ένα συγκεκριμένο χώρο. Αυτό νομίζω η κυρία Μπρέσο το καθιστά απόλυτα σαφές στην προσέγγιση που υιοθετεί. Αλλά πρέπει να προσέξουμε όταν λέμε για διάθεση πρόσθετων κονδυλίων, γιατί αυτό δύσκολα θα επιτευχθεί και θα μας δυσκολέψει και στη δικιά μας τη δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς στην τελική διατύπωση του κειμένου στην έκθεση, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι ε, θα γίνουμε σωστά κατανοητοί. Ο κύριος Μπόγκοβιτς είναι ο επόμενος ομιλητής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να συγχαρώ την κυρία Μπρέσο. Η έκθεση είναι εξαιρετική. Ε, αναφέρεται στις μακροπεριφέρειες, στην τέταρτη μακροπεριφέρεια. Όπως είπε η κυρία Μπρέσο, αυτή είναι η πρώτη στρατηγική η οποία εστιάζει σε ορεινές περιοχές, σε μια ορεινή περιοχή. Πάντα μας απασχολούν τα κονδύλια όταν μιλάμε για τέτοιες στρατηγικές, αλλά εγώ είμαι πεπισμένος ότι είναι σημαντικό να προωθήσουμε τη συνεργασία των κατοίκων αυτών των περιοχών, διότι αυτές οι περιοχές επλήγησαν από πολέμους, τον πρώτο, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και οπωσδήποτε ε, υπέστησαν συνέπειες όταν μιλάμε για μακροπεριφέρειες, είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας και την προσφυγική κρίση. Ε, αυτό ενδιαφέρει πολύ την Ιταλία-Αυστρία. Γι' αυτό τονίζω ότι αυτή η μακροστρατηγική σημαίνει κάτι πολύ παραπάνω από μια συζήτηση για τους χρηματοοικονομικούς πόρους. Όπως είπατε, μιλάμε για 80 εκατομμύρια ανθρώπους που μεταξύ άλλων ζουν και σε πολύ απομονωμένες ορεινές περιοχές. Ε, αλλά και ε, το, πρόβλημα τότε το αντιμετωπίζουν και οι άνθρωποι που ζουν στις πόλεις. Πρόκειται λοιπόν για συνεργασία μεταξύ των παιδινών και ορεινών περιοχών. Επίσης πρέπει να γνωρίζουμε ότι η περιοχή αυτή έχει επίδραση σε ολόκληρη την Ευρώπη σε ό,τι αφορά την ε, παροχή ίδρευσης, για παράδειγμα. Οι τρεις πυλώνες είναι, κατά τη γνώμη μου, σωστοί η ανταγωνιστικότητα και η καινοτομία είναι πολύ σημαντικό τομέας, πολύ σημαντική περιοχή αυτή με πολλές καινοτομίε και ισχυρή οικονομία στις παιδιάδες. Στις ορεινές περιοχές πρέπει να μας απασχολήσει η προστασία της φύσης, ο τουρισμός και η κτηνοτροφία. Η γεωργία κτηνοτροφία. Αν δεν υπάρχει οικονομία στις ορεινές περιοχές, δεν θα υπάρχουν δυνατότητες επιβίωσης. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντική η ανάπτυξη αυτών των περιοχών. Η κινητικότητα, η διασύνδεση είναι πράγματα σημαντικά βεβαίως. Οι, οι σιδηρόδρομοι, οι μεταφορές εμπορευμάτων, η μεταφορά των, ε, από τις ε, οδικές τις ιδροδρομικές μεταφορές, το πέρασμα, οι ψηφιακές διασυνδέσεις, οι μεταφορικές διασυνδέσεις με τις ορεινές περιοχές, το περιβάλλον, η ενέργεια, όλα αυτά είναι σημαντικά. Η κλιματική αλλαγή επίσης, όλα παίζουν μεγάλο ρόλο. Είδαμε τώρα ότι υπάρχουν πολλές πλημμύρες λόγω του, των ήπιων χειμώνων που προηγήθηκαν. Αυτό αλλάζει την ε, κατάσταση και το ισοζύγιο των υδάτων. Επίσης υπάρχουν σημαντικές πηγές ενέργειας, αιωλική, ηλιακή. Και όλα αυτά είναι σημαντικά αφού και ε, ε, εδώ υπάρχει διαφορετικός ενεργειακός εφοδιασμός οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι πολύ σημαντικές. Έγινε στις 25-26 Ιανουαρίου μια πρώτη ε, διάσκεψη στη Σλοβενία και χάρηκα πρέπει να πω διότι συγκεντρώθηκαν 400 σύνευροι από πολλές περιοχές, πολλές πόλεις και δημιουργήθηκε μια δομή διοίκησης θα γίνει και σήμερα μια συνάντηση στο Κούσελστατ. Το Φεβρουάριο θα έχει κλείσει μια εικοσαετία από τη σύμβαση, την έγκριση της σύμβασης των Άλπαιων και είμαι πεπισμένος ότι αυτή η μακροστρατηγική θα είναι πολύ επιτυχής. Είμαι πεπισμένος επίσης ότι θα μας απασχολήσουν και άλλα θέματα και όχι μόνο για τα ευρωπαϊκά, κονδύλια. Είναι σημαντικό να έχουμε συμπράξει όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Αν δεν θέλει κανείς άλλος το λόγο, θα δώσω το λόγο στην κυρία Φιλομένα Καρλάνου, που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μπρέσο καταρχήν για την εξαιρετική της έκθεση και για τις συστάσεις της, τις ε, οποίες συμμεριζόμαστε σχεδόν στο σύνολό τους. Ε, τρία σημεία υπογραμμίζονται που πιστεύω ότι είναι και τα πιο σημαντικά. Πρώτον, το θέμα της ε, διακυβέρνησης στρατηγικής, ε, το θέμα της χρηματοδότησης και το ζήτημα της ε, διάρθρωσης γιατί για πρώτη φορά πρόκειται για μια στρατηγική που δεν αφορά μόνο ορεινές περιοχές, ορεινούς όγκους, αλλά και όλες τις ε, γύρω περιοχές ε, που περιβάλλουν τον ορεινό όγκο. Πρόκειται λοιπόν για μια ολοκληρωμένη σφαιρική στρατηγική που αφορά μια οροσυρά και παιδιάδες γύρω από αυτήν. Η Κομισιόν αναγνωρίζει την ευθύνη της και είναι πρόθυμη να παίξει ρόλο στο στρατηγικό συντονισμό. Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω ότι αυτή η στρατηγική είναι προϊόν, αποτέλεσμα μιας ε, ισχυρής επιθυμίας ε, συγκεκριμένων χωρών που συμμετέχουν σε αυτή την περιφέρεια. Οπότε, ε, είναι σημαντικό και αυτές οι χώρες κάθε μία στο εσωτερικό της ε, να θέσει στη διάθεση της στατικής αυτής επαρκής πόρους και ανθρώπινο δυναμικό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει να παίξει επίσης ε, σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση της στρατηγικής. Οπότε πρέπει, μάλλον η πρόταση του Κοινοβούλιο να συμμετάσχει στη διακυβέρνηση είναι πολύ καλή. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση της ε, στρατηγικής, μιλούμε για δύο διαφορετικούς τύπους χρηματοδότησης. Πρώτον, χρηματοδότηση σχεδίων. Η στρατηγική αυτή δεν είναι ένα καινούριο πρόγραμμα που θα χρηματοδοτηθεί από τα διευθυντικά ταμεία. Η ίδια στρατηγική δεν διαθέτει πόρους σε Οπότε αυτό που θα πρέπει να παίξει, αυτό, αυτό, θα πρέπει να είναι ο ρόλος της, είναι ο συντονισμός Έχουμε πάνω από 80 προγράμματα τα οποία παρεμβαίνουν στην ίδια ζώνη, στην ίδια περιοχή, οπότε η στρατηγική θα συντονίσει όλα αυτά τα προγράμματα, θα τα διαρθρώσει και θα τους δώσει και στρατηγικό χαρακτήρα. Πώς, ε, είτε με προσκλήσεις ενδιαφέροντος για συγκεκριμένα σχέδια, ε, με προτεραιότητες σύμφωνες με τις προτεραιότητες της στρατηγικής, ε, ο στόχος είναι προγράμματα τα οποία ήδη είναι ανοιχτά και λειτουργούν να συνεισφέρουν στους στόχους της στρατηγικής. Μετά, έχουμε και τη χρηματοδότηση της ίδιας διακυβέρνησης στρατηγικής. Και εκεί ε, έχουμε το εξή ε, φαινόμενο. Έχουμε το Alpine Space, ε, που είναι ένα πρόγραμμα που θα πρέπει να στηρίξει διοικητικά τη στρατηγική, αλλά οι πόροι του είναι περιορισμένοι, οπότε συστήνουμε το Κοινοβούλιο, όπως έκανε και με τις άλλες τρεις προηγούμενες στρατηγικές, να ε, διαθέσει πόρους από τον ίδιο το δικό του προϋπολογισμό, για παράδειγμα για τη χρηματοδότηση μελετών ε, ή για κονδύλια έναρξης, ε, seed money όπως λέγεται κλπ. Σε ό,τι αφορά τους θεματικούς στόχους, η στρατηγική έχει τρεις θεματικούς στόχους, αλλά υφίσταται και ένας τέταρτος στόχος που είναι οριζόντιος, δεν είναι θεματικός και είναι η διακυβέρνηση. Με τον αριθμό των δομών και οργανώσεων που υπάρχουν ήδη στην περιοχή αυτή, πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό όλες αυτές οι δομές να διαρθρωθούν σωστά έτσι ώστε να αποφύγουμε τις αλληλεπικαλύψεις και να δώσουμε νόημα σε όλες τις παρεμβάσεις που ήδη γίνονται. Ευχαριστώ. Thank you. Thank you very much. Ευχαριστώ. Κύριε Μπρέσο, θέλετε να ολοκληρώσετε τη σημερινή μας συζήτηση. Ευχαριστώ. Πολύ άριθμες οι παρατηρήσεις. Ορισμένες μάλιστα μπαίνουν σε μεγαλύτερες λεπτομέρειες και μπορούμε να τις συζητήσουμε στη συνεδρίαση των σκιωδών. Εγώ θέλω να μιλήσω για κάποιες παρατηρήσεις κλειδιά που ακούστηκαν σε αυτή τη συζήτηση. Πρώτη, το θέμα της χρηματοδότησης. Μας υπενθυμίσατε ότι δεν θέλουμε επιπρόσθετες ε, χρηματοδοτήσεις αλλά ότι η πολιτική συνοχής, η οποία έχει πάρα πολλούς πόρους για αυτή την περιοχή, θα πρέπει να επιτύχει τη σύγκληση όλων αυτών των πόρων γύρω από τους στρατηγικούς στόχους. Κάτι που, όπως υπενθύμησε και εκπρόσωπος της Κομισιόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποφύγουμε τον κατακαιρματισμό ή την αλληλεπικάλυψη των project, των έργων. Οι περιφέρειες και οι τοπικοί φορείς, οι οποίοι θα πάρουν στα χέρια τους αυτή την διακυβέρνηση της στρατηγικής, την governance με συγκεκριμένους όρους στρατηγικής, θα πρέπει να διαθέσουν και ανθρώπινους και οργανωτικούς πόρους για να εξασφαλιστεί ένα σωστός συντονισμός. Τόσο να υπάρχει μια ενσωμάτωση ολόκληρη, μια ένταξη ε, σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, ενιαίο πλαίσιο όλης της αλπικής περιοχής. Τώρα, με την ανάπτυξη των μακροπεριφερειακών στρατηγικών μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, καθώς και το σχέδιο Juncker. Ίσως υπάρξουν και, άλλες, ε, και άλλα έργα ε, και μπορούμε χάρη σε αυτά τα λεφτά να βοηθήσουμε τους τοπικούς φορείς ούτως ώστε να δημιουργηθούν πλατφόρμες χρηματοδότησης, όχι επιπλέον κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πλατφόρμες ούτως ώστε να μπορέσουν να ελκύσουν επενδύσεις και από τον τραπεζικό τομέα αλλά και από δημόσιους, ε, συγγνώμη, ιδιωτικούς επενδυτές. Επ' αυτού σκεφτήκαμε, εργαστήκαμε, μιλήσαμε και θα το συζητήσουμε ξανά στη συνεδρίαση των σκιωδών. Εγώ πιστεύω ότι για τα στρατηγικά θέματα για την Ευρώπη και για τον κόσμο, όπως η βιοπικιλότητα, η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η δυνατότητα να έχουμε πειραματικά project, Παραδείγματο χάρη για την κυκλική οικονομία, όπως υπενθύμισε ο συνάδελφος αυτή την περιοχή, μπορούμε εκεί να χρησιμοποιήσουμε διάφορα άλλα κονδύλια ευρωπαϊκά που δεν θα αφορούν τη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά κάποια θέματα που αφορούν την περιοχή εν συνεχεία μπορεί να υπάρξει και συμμετοχή και άλλων τμήματων της Ευρώπης, είτε ορεινών ή μη, που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά. Αν έχουμε όμως ε, κονδύλια από το Horizon, από το COSME, από διάφορα, διάφορα προγράμματα, οι πόρους, οι εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το LIFE κτλ. που θα μας επιτρέπουν να αντιμετωπίσουμε κάποια από τα μεγάλα θέματα, τα, τις μεγάλες ερωτήσεις, τις κρίσιμες ερωτήσεις που με τις οποίες ασχολείται και αυτή η στρατηγική, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όταν λέμε λοιπόν χρηματοδότηση, δεν εννοούμε νέα χρηματοδότηση. Τη δυνατότητα να προσανατολίσουμε τους πόρους, δημόσιους και ιδιωτικούς, προς τη σωστή κατεύθυνση μέσω αυτών των ειδικών τόπων ή πλα... ονομάζουμε πλατφόρμες ε, επένδυσης. Ευχαριστώ την Κομισιόν που εκτιμάει την προσπάθεια του Κοινοβουλίου για να παρεμβαίνει πιο συγκεκριμένα στα θέματα της governance, που είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο της ε, αυτοοργάνωσης της περιοχής. Είναι σημαντικό να συμμετέχουμε και να είμαστε παρόντες, ούτω ώστε να καταλάβουμε καλύτερα ως ε, νομοθέτες τις ανάγκες που έχουν οι διάφορες ε, περιοχές. Και δεν μιλάμε μόνο για την αλπική περιοχή, για πολλές περιοχές που οργανώνονται με βάση την αρχή της εδαφικής συνοχής, οργανώνονται λοιπόν για να εκμεταλλευθούν καλύτερα το δυναμικό που προσφέρει και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αλλά και η Ευρωπαϊκή Πόρη. Για το θέμα των μεταφορών. Συμφωνώ με πάρα πολλές από τις παρεμβάσεις που άκουσα Πέρα από τη στρατηγική υπάρχουν ε, τα λεγόμενα ε, τα διευρωπαϊκά δίκτυα για τις μεταφορές, που έχουν εγκριθεί, χρημα, ε, υπάρχει χρηματοδότηση κτλ. Για να υποφεληθεί η περιοχή αυτή από αυτές τις επενδύσεις, από αυτά τα έργα δηλαδή, πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη διασύνδεση όλης της περιοχής, δηλαδή της αλπικής, καθ' αυτό αλπικής, αλλά και της περιαλπικής. Και το υπενθύμησαν πολλοί συνάδελφοι. Η δυσκολία των διασυνδέσεων. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε όλες τις ευκαιρίες. Και αυτό είναι το στρατηγικό σημείο για τη μακροπεριφέρεια. Η διασύνδεση. Που έχει αυτές τις μεγάλες διασυνδέσεις, τους μεγάλους άξονες, αλλά που κινδυνεύουν να την αφήσουν έξω. Δηλαδή θα υπάρχουν μεν οι άξονες, αλλά δεν θα συνδέουν πραγματικά ολόκληρη την περιοχή και τις διάφορες υποπεριοχές. Τώρα, το θέμα της governance είναι να μην αφήσουμε μόνες αυτές τις περιεφέρειες, τις περιοχές. Η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο, τα κράτη προφανώς, θα πρέπει να ασχοληθούν. Αλλά θα πρέπει οι ίδιες οι περιοχές αυτές να αφυπνιστούν, να υπάρξει μια επίγνωση η περιοχή αυτή δεν είναι ούτε καθ' αυτό ορεινή, ούτε μόνο, παιδινή, ούτε μόνο ορεινή, ούτε μόνο παιδινή. Για πρώτη φορά υπάρχει ένας διάλογος ανάμεσα στις ορεινές και παιδινές περιοχές. Και θα πρέπει και οι δύο να υποφεληθούν από τον προγραμματισμό, από τη χρηματοδότηση κτλ. Αλλά η governance των περιφερειών αυτών, των περιοχών, είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί προκύπτουν διάφορα συγκεκριμένα έργα, άρα χρειαζόμαστε συντονισμό. Εδώ μιλάμε για μια περιοχή όπου Όλες οι περιφέρειες, ε, υποπεριφέρειες δηλαδή των, της μακροπεριφέρειας αυτής, έχουν νομοθετικές εξουσίες και εκείνες διαχειρίζονται τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής. Επομένως, αυτές οι περιφέρειες θα πρέπει να δείξουν ότι έχουν τη δυνατότητα να φτιάξουν την αποτελεσματική αυτή governance που καταφέρνει να εξασφαλίσει την υλοποίηση των στόχων. Και μιλάμε για μια στρατηγική που για πρώτη φορά γεννήθηκε από, τα, από, από κάτω, από τη βάση. Είναι μια στρατηγική bottom-up. Θα πρέπει αυτή η δυνατότητα governance να δείξει ότι έχει δυνατότητα ε, να παράγει απτά έργα. Ακούστηκαν πάρα πολλά πράγματα και φυσικά θα ενταχθούν μέσω των τροπολογιών καθώς αρχίσω να τα σκέφτομαι, ε, να ξανασκέφτομαι την έκθεσή μου, θα λάβω υπόψη προφανώς πολλά από τα θέματα που θέσατε. Έχω, τα έχω σημειώσει, επιμελώς. Καταληκτικά. Μπορούμε να το συζητήσουμε το θέμα της governance και με την Κομισιόν. Πώς μπορούμε να την ξαναδούμε, να την ξαναφανταστούμε, να την ξαναφτιάξουμε, ούτως ώστε να εντάξουμε καλύτερα το Κοινοβούλιο σε όλο αυτό το μηχανισμό. αυτή η συμμετοχή του Κοινοβουλίου είναι καλή ε, και για αυτή τη στρατηγική των Άλπων, αλλά και, για άλλε στρατηγικέ μελλοντικέ ενδεχομένω. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπρέσο. Θυμίζω στου συναδέλφου ότι η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι 3η 26 Απριλίου στις 5 το απόγευμα. Στη συνά... Και την Τρίτη στις 9 είναι η συνάντηση των σκιωδών. Εντάξει. Τρίτη σκιώδης, προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών την είπαμε. Τρίτη, 26 Απριλίου. Λοιπόν, Ολοκληρώσαμε τη συζήτηση για αυτό το σημείο τη ημερήσιας διάταξης και συνεχίζουμε με μια ανταλλαγή απόψεων με την κυρία Λίζα Μπόνη, Γενική Γραμματέα της EuroCities. Πού είναι η προσκεκλημένη μας. Ήρθε. Στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος ελέγχου ε, καλέσαμε τις EuroCities για ανταλλαγή απόψεων σε πολλά θέματα, κυρίως την αστική διάσταση της πολιτικής συνοχής. Η EuroCities είναι η φωνή των ευρωπαϊκών πόλεων στις Βρυξέλλες, περιλαμβάνει μεγάλες πόλεις, που έχουν εκλεγεί με τοπική δημοτική κυβέρνηση μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Η οργάνωση συνδυάζει τοπικές κυβερνήσεις του ΣΟΤΑ, δηλαδή 130 από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ευρώπης και 40 ε, πόλεις που ε, εκπροσωπούν πάνω από 130 εκατομμύρια ε, ε, κατοίκους από 35 χώρες. Ε, έχουμε πολλά συστηματικά φόρουμα, ομάδες εργασίας, δραστηριότητες, εκδηλώσεις και έτσι η EuroCities προσφέρει μια πλατφόρμα ε, διαμοιρασμού γνώσης και ανταλλαγής ε, εμπειριών. Τα EuroCities έχουν εκφράσει ισχυρή υποστήριξη μιας πολιτικής χωρίς αποκλεισμούς ανοιχτές σε όλες τις περιφέρειες και τις πόλεις για να αντιμετωπιστούν τωρινέ και μελλοντικέ προκλήσεις στην Ευρώπη με μετροπολιτική εστίαση και ολοκληρωμένη πολιτική που θα στηρίζεται σε συμπράξει γνήσιε. Η κυρία Άννα Ελίζα Μπόν, Γενική Γραμματέας της Γιουροσίτη, ήρθε εδώ σήμερα για να παρουσιάσει ορισμένες από τις σημαντικότερες προτεραιότητες που θέλουν οι Γιουροσίτη στην πολιτική συνοχής με ιδιαίτερη εστίαση και πέραν του 2020 ίσως. Αλλά μπορείτε βεβαίως να μας πείτε ό,τι έχετε ε, επιλέξει να μοιραστείτε μαζί μας. Έχετε το λόγο κυρία Άννα Λιζαμπόνη. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ που καλέσατε τις EuroCities να ε, εκφράσουν τις απόψεις τους εδώ. Πολλοί μας γνωρίζετε ήδη γιατί έχουμε ήδη παρέμβει ιδιαίτερα στο θεματολόγιο για τις πόλεις. Ευχαριστούμε λοιπόν και χαιρετίζουμε το ενδιαφέρον των μελών της Επιτροπής σας, της Επιτροπής ε, Ρέτζι, που θέλετε να ακούσετε τι θα πούμε τώρα και για την επόμενη περίοδο. Καλό είναι να αρχίσω με μια σύντομη αναφορά στην ε, urban agendas, δηλαδή στο θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πόλεις, αστικό θεματολόγιο, γιατί βλέπω και τον εισηγητή που είχε ασχοληθεί με το θέμα, κάνατε και εσείς συζητήσεις, να δώσω κάποια μηνύματα για το πώς θεωρούμε ότι θα κινηθούν τα πράγματα προς το Άμστερνταμ και το σύμφωνο του Άμστερνταμ. Προϋποθέτω ότι τη διαδικασία την ξέρετε αφού ήρθε και σας μίλησε και η Ολλανδική Προεδρία, αλλά και το τι θα γίνει μετά το Άμστερνταμ. Κάποια κέρια λοιπόν μηνύματα και θέματα. Για μας το κείμενο ως έχει σήμερα το σχέδιο συμφώνου του Άμστερνταμ είναι ένα αποτέλεσμα καλό. Μιλώντας γενικά, γιατί ήταν ε, τα προηγούμενα 20 χρόνια στο στόχαστρο των συζητήσεων και με βάση αυτό κρίνουμε ότι είναι καλό γιατί είναι πολύ πιο συγκεκριμένο από ό,τι ήταν στο παρελθόν που ακούγαμε πολλές δηλώσεις, διακηρύξεις κλπ. Πάει στη σωστή κατεύθυνση. Και πρώτη φορά τα κράτη-μέλη είναι έτοιμα να παίξουν το παιχνίδι συλλογικά γύρω από τον αστικό χώρο. Ίσως γιατί δεν φοβούνται πια ότι εμείς πιέζουμε προς την κατεύθυνση μιας πολιτικής. Γιατί αυτή, αυτό το ενδεχόμενο τους ανησυχεί σε ό,τι αφορά επικουρικότητα κλπ. Πρέπει να πω ότι η έκθεσή σας συν η Ολλανδική Προεδρία η οποία ε, έδωσε μεγάλη όθηση σε αυτή την πρωτοβουλία αλλά και η τωρινή προσπάθεια της Γενικής Διεύθυνσης θέλω δηλαδή την ε, μονάδα για τις πόλεις πρέπει να τη συγχαρώ έπαιξε μεγάλο ρόλο για να ε, προχωρήσει η συζήτηση οπότε αυτά είναι καλά υπόσχονται πολλά οι σημερινές εξελίξεις αλλά θα προσθέσω κάποια σημεία το σύμφωνο το χρειαζόμαστε για να διασφαλίσουμε την παροχή συγκεκριμένων δράσεων. Πρέπει να υπάρχει σαφής αντίκτυπος του θεματολογίου, δηλαδή να βελτιωθεί η ζωή της πόλης. Αν δεν το εξασφαλίσουμε αυτό, τότε δουλεύουμε ματέως. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μηχανισμούς παράδοσης όπως οι συμπράξεις, οι εταιρικέ σχέσεις, τα προγράμματα δράσης και η, παροχή τους, η παράδοσή τους θα πρέπει να διέπονται από την ανάγκη επίλυσης των προβλημάτων που θέτουν επιτάπητος οι πόλεις. Δεν πρέπει να προέρχονται δηλαδή τα θέματα αυτά από τα κράτη-μέλη αλλά από τις πόλεις τις ίδιες. Δείτε το προσφυγικό. Δεν ξέρω αν είδατε την έκθεση που καταρτήσαμε πρόσφατα ε, καταγράφουμε ανάγκες, τάσεις, πράγματα που συμβαίνουν στις πόλεις. Αν υπάρχει θεματολόγιο λοιπόν πόλεων πρέπει να διέπεται από τις ανάγκες αυτές. Πρέπει να βοηθήσουμε να βελτιωθεί η πολιτική και οι κανονισμοί για τις πόλεις. Αυτό είναι μεγάλο κομμάτι. Δηλαδή το θεματολόγιο για την καλύτερη νομοθεσία θα πρέπει σαφώς να συνδέεται στο θεματολόγιο για τις πόλεις και αντίστροφα. Οι μηχανισμοί παράδοσης όπως ε, μελέτες επιπτώσεων που θα πρέπει να υπάρχουν επιτάπητος γιατί εντάσσουν τις πόλεις σε μία ε, εκ των προτέρων αναθεώρηση ή εξέλιξη της πολιτικής και έτσι ο κανονισμός θα έχει καλύτερο αντίκτυπο επιτόπου. Ε, υπάρχουν πολλά παραδείγματα εδώ, στέγαση, ποιότητα της ατμόσφαιρας, πρόσφυγες, μετανάστες, ενσωμάτωση κλπ. Και μπορεί να πάει, να βοηθήσουν να πάει η χρηματοδότηση στο σωστό στόχο. Σήμερα δεν είναι εύκολο αυτό. Δεν πάνε τα λεφτά εκεί που πρέπει πάντα. Σε πολλές περιπτώσεις μπλοκάρονται στο εθνικό επίπεδο. Αυτό λοιπόν ήταν η πρώτη μου παρατήρηση, πολύ συγκεκριμένα. Δεύτερον, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η 30η Μαΐου δεν θα είναι το τέλος μιας διαδικασίας, αλλά η αρχή μιας νέας διαδικασίας, ακόμα πιο σημαντικής. Όταν παραδώσουν οι Ολλανδοί, τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε μετά τους Ολλανδούς. Ε, ως Προεδρία εννοώ να παραδώσει. Αυτό που ζητούμε είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ενισχυθεί σε αυτή τη συντονιστική διαδικασία, να διατεθούν οι σωστοί πόροι, να αναλάβουν όλοι τα πολιτικά αυτά προγράμματα στο επίπεδο που πρέπει και να τα οικειοποιηθούν. Ένα σημαντικό στόχος είναι η καλύτερη νομοθεσία, ο καλύτερος συντονισμός, ε, κοινή ε, ενωσιακή πολιτική. Αυτός είναι θεμητό στόχος και θέλουμε την άποψή σα επί όλων αυτών. Επί όλων Τρίτον, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι πόλεις θα συμβάλλουν σε μηχανισμούς όπως συμπράξεις, εταιρικές σχέσεις και δεν θα είναι μεμονωμένες φωνές, γιατί έτσι είναι σήμερα η κατάσταση. Ίσως η απόσταση είναι μεγάλη από τις πόλεις μέχρι εσάς. Οι πόλεις θέλουν να ενταχθούν στις συμπράξεις με εκπροσώπηση κλπ. Το σημαντικό εδώ είναι να διασφαλίσουμε ότι τα μηνύματα που κατατίθενται σε αυτό το τραπέζι θα είναι μηνύματα που αφορούν το συνολικό αστικό σύστημα, το σύστημα των πόλεων εννοώ. Αν πάρουμε ας πούμε την προσφυγική κρίση, αν υπάρχουν πόλεις γύρω από το τραπέζι που δεν θα λένε μόνο «Α, ε, θέλουμε να είμαστε εδώ» ή «Αυτή η πόλη θέλει να πάει εκεί» είτε πρόκειται για τη λειψία ή το μόναχο κλπ. Όχι. Όχι με μονομένη προσέγγιση. Θα πρέπει τα βασικά σημεία να μπουν στο τραπέζι. Ο ρόλος των πόλεων θα πρέπει να αναγνωριστεί δηλαδή στους επόμενους κανονισμούς που θα διέπουν αυτή την πολιτική, ότι θα είναι σωστή η χρηματοδότηση, ώστε για παράδειγμα το ε, πρόγραμμα και η χρηματοδότηση για την ενσωμάτωση των προσφύγων να είναι διασφαλισμένα, τέτοια πράγματα. Και εδώ βέβαια χρειάζονται ενώσεις όπως η δική μας, γιατί και μας αυτό μας απασχολεί, να έχουμε ένα θεσμικό πλαίσιο σε τελευταία ανάλυση για να αξιοποιήσουμε τα μηνύματα που στέλνουν οι πόλεις. Εδώ και χρόνια για την ποιότητα της ατμόσφαιρας το είπαμε και το ξανά είπαμε ότι χρειαζόμαστε πολύ πιο συντονισμένη πολιτική μεταξύ Γενικής Διεύθυνσης, ε, Περιβάλλοντος, Κλίματος και άλλες ε, διευθύνσεις. Δεν ε, θέλουμε μία μεμονωμένη πόλη ή μια άλλη πόλη από μόνη της. Θέλουμε να πούμε ότι αυτά το κράτος μέλος, οι Κομισιόν κάνουν για τη συμφόρηση τα τάδε πράγματα για να συμβάλλουμε στην ποιότητα της ατμόσφαιρας π.χ. της πόλης. Πρέπει λοιπόν να είναι βέβαιο ότι θα υπάρχουν εκπρόσωποι των σωστών οργανώσεων ε, θα βρίσκονται γύρω από το τραπέζι μαζί με την ομάδα παρακολούθησης από τη Γενική Διεύθυνση. Δεν θα είμαστε μόνο παρατηρητές βεβαίως, αλλά θα παίζουμε ρόλο, θα παρεμβαίνουμε. Με αυτές τις συμπράξεις δεν πρέπει να δημιουργηθούν καινούργιοι βαρύς μηχανισμοί, γιατί αυτό ενέχει κίνδυνο να δαπανηθούν ε, χρήματα σε συναντήσεις ε, και μόνο. Ενώ ήδη συμβαίνουν πολλά ε, μέσα από δίκτυα όπως το δικό μας και όχι μόνο. Δίκτυα στα κράτη-μέλη, στις ε, γενικές διευθύνσεις κλπ. Πρέπει όλα αυτά να τα αξιοποιήσουμε. Αν χρειάζεται σύμπραξη για την ε, ποιότητα της ατμόσφαιρας, είχαμε ωραίο παράδειγμα. Την περασμένη εβδομάδα έγινε ένα δίκτυο το, για το περιβάλλον, 56 πόλεις ε, ήρθαν σε επαφή με τους σωστούς ανθρώπους, με τις γενικές διευθύνσεις, την Κομισιόν κλπ. Ε, τώρα οι πόλεις δεν έχουν πόρους ε, να δαπανούν ε, για συμμετοχή σε συναντήσεις και μόνο. Θα πρέπει να υπάρχει σαφές αποτέλεσμα από όλα αυτά. Αυτό λοιπόν είναι ένα μήνυμα που θα ήθελα εγώ να Φέρω εδώ, σε αυτό το χώρο. Τέλος. Για τα κράτη-μέλη και πάλι, είδαμε ότι σε αυτές τις συμπράξεις ή τις εταιρικέ σχέσεις δεν συμμετέχουν πολλοί. Η Κομισιόν παίζει το παιχνίδι, όπως σας είπα, αλλά από τα κράτη-μέλη όχι. Έχουμε ένα, δύο ανά εταιρική σχέση. Αν θέλουμε να ε, αντιμετωπίσουμε τη συμφόρηση και να έχουμε καλύτερη νομοθεσία, πολλοί φραγμοί προσκόμματα της νομοθεσίας ε, παρατηρούνται σε εθνικό επίπεδο. Ως ε, Ευρωβουλευτές λοιπόν, ως Επιτροπή υπεύθυνη για το θεματολόγιο για τις πόλεις, τι μπορείτε να κάνετε, τι άποψη έχετε και τι μπορείτε να συνεισφέρετε στο εθνικό επίπεδο για να αυξηθεί η συμμετοχή των κρατών μελών και να παίξουν το παιχνίδι. Όχι σε εθνικό επίπεδο, αλλά συνολικά στα πλαίσια του θεματολογίου για τις πόλεις επίσης, να παίξουν το ρόλο των πολλαπλασιαστών. Και αυτός είναι ένας ρόλος τους για να φτάσει το θεματολόγιο για τις πόλεις μέχρι τη βάση, μέχρι το συνολικό σύστημα των πόλεων σε κάθε κράτος μέλος. Αυτά πρέπει να γίνουν το ταχύτερο δυνατόν και αυτά ήταν αυτά που είχα να πω όσο γίνεται πιο γρήγορα ως βασικά θέματα προκειμένου να έχω μια ανταλλαγή απόψεων μαζί σας για το θεματολόγιο των πόλεων. Αν έχετε ερωτήσεις ευχαρίστω να απαντήσω γιατί έχουμε και την πολιτική συνοχή. Μπορούμε και αυτή να τη συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ήδη έχουμε ένα σύντομο κατάλογο μιλητών. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, Αναλύζα ε, Πολλές φορές ε, συναντηθήκαμε μαζί να μιλήσουμε και για το θεματολόγιο των πόλεων και μετά συναντηθήκαμε και διαπιστώνω ότι προφανώς επιλέξαμε τη σωστή στιγμή για την έκθεση. Όλα αυτά που μας είπες μόλις τώρα ε, εκτίμηση επιπτώσεων, χρηματοδότηση, εταιρικέ σχέσεις ή συμπράξεις, όλα αυτά υπάρχουν και στην έκθεση γιατί επιτέλους θέλουμε να τελειώσουν αυτές οι πολιτικές ε, οι, ε, για τις πόλεις. Πρέπει να είναι στοχοθετημένες. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει με τις συμπράξεις ή τις εταιρικέ σχέσεις, τα partnerships αυτά. Από ό,τι γνωρίζω εγώ, εδώ μεταξύ υπάρχουν πέντε τέτοιες συμπράξεις και στο, για το προσφυγικό, για την ε, ε, φτώχεια στις πόλεις, για τη στέγαση και 15 άνθρωποι συμμετέχουν σε αυτές τις συμπράξεις και από, από εσά αλλά και από άλλες οργανώσεις. Τελευταία, ε, μίλησα με την Ένωση Δήμων στη Γερμανία, γιατί είπες ότι στις 30 Μαΐου δεν τελειώνει το θεματολόγιο, αντίθετα μάλιστα. Πρέπει να προχωρήσουμε, γιατί τότε θα έχουμε πραγματικές επιτυχίες. Μόνο και μόνο το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο και η Προεδρία της Ολλανδίας συνεργάζεται καλά με τις πόλεις, και μάλιστα στο σύμφωνο του Άμστερνταμ υπάρχουν ορισμένα πράγματα που πρέπει να διορθωθούν. Δεν συμφωνούμε με όλα, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο, όπως είπες και εσύ. Όμως και πέρα από όλα αυτά πρέπει να γίνει μια σωστή δουλειά. Νομίζω ότι η Κομισιόν τώρα ε, έχει μπει στο παιχνίδι, δημιούργησε αυτές τις συμπράξεις, δεν θα είναι οι μοναδικές, ε, ε, θα έχουν διάρκεια τριετή και στο τέλο θα πρέπει να έχει επιτευχθεί ένα στόχος, να έχει βγει ένα αποτέλεσμα το οποίο θα το εφαρμόσουν οι πόλεις και όχι μόνο οι μεγαλοπόλεις αλλά και οι μικρομεσαίες πόλεις, οι λειτουργικοί χώροι, όλα αυτά είναι γνωστά και υπάρχουν και στην έκθεση. Και η Γερμανική Ένωση Δήμων ενδιαφέρθηκε πάρα πολύ, έχει κάνει δημοσιεύσεις παντού Βέβαια, καμιά φορά υπάρχουν δυσκολίες να πιστούν οι πόλεις να συμμετέχουν σε αυτές τις συμπράξεις. Γιατί όντως δεν ξέρουν πολύ καλά τι ικανότητες πρέπει να διατεθούν ακριβώς. Και εδώ ίσως θα χρειαστούν κάποιες διευκρινήσεις για την Κομισιόν θα πρέπει να γίνει δικτύωση, η μελέτη επιπτώσεων, τι κάνουν οι διάφοροι τομείς. Αυτό είναι νερό στο μήλο μας. Ε, εμείς έτσι το έχουμε διατυπώσει το θέμα όταν είπαμε ότι θέλουμε σε υψηλό επίπεδο έναν συντονισμό. Για να δούμε αν, θα, αν αυτά θα ε, καταγραφούν σωστά και στο σύμφωνο του Άμστερνταμ. Ευχαριστώ πολύ και επαναλαμβάνω δεν τελειώνουν όλα στις 30 Μαΐου. Ίσα ίσα θα πρέπει να γίνει μια νέα αρχή τότε. Ευχαριστώ κυρία Μαλεβίτς. Ευχαριστούμε πολύ για την εισαγωγή σας κυρία Μπόνη. Υπογραμμίσατε κάτι πολύ σημαντικό που έχει σχέση με την εφαρμογή του θεματολογίου για τις πόλεις. Είπατε ότι συμμετέχει το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή, ε, οι πόλεις, αλλά λείπουν τα κράτη-μέλη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πώς είναι δυνατόν να υλοποιηθεί το θεματολόγιο για τις πόλεις χωρίς τη συμμετοχή των κρατών μελών. Πρέπει να στηρίξουν τις πόλεις και να τις εναρμονίσουν έχουμε και οριζόντια, πολλά οριζόντια θέματα, αλλά και ε, τομεακά. Και εκεί θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις σε συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια για τις Εθνικές Κυβερνήσεις. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσαμε να διευκολύνουμε τις συζητήσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια σε ό,τι αφορά την ε, συζήτηση της υλοποίηση του θεματολογίου για τις πόλεις. Γιατί χρειάζεται τα Εθνικά Κοινοβούλια και τα συναρμόδια Υπουργεία να συνεισφέρουν ενεργά στην υλοποίηση του θεματολογίου σε εθνικό επίπεδο. Ευχαριστώ και ο Σόλμπρεχτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Γνωρίζουμε τις δραστηριότητες του δικτύου EuroCities. Ξέρουμε πόσο ισχυρή είναι η επίδραση του δικτύου η Ολλανδική Προεδρία πρότεινε την εταιρική σχέση, ε, μια μορφή η οποία ήδη υπάρχει μεταξύ των πόλεων. Η ανταλλαγή εμπειριών αφορά όχι μόνο το παρελθόν, αλλά και την ε, εργασία για τη μελλοντική δράση. Οπότε είναι σημαντικό που αυτό, αυτή η μορφή συνεργασίας μετακφέρεται σε άλλο επίπεδο πλέον. Αυτό το μείγμα των 15 που είναι μυρογνώμονες, οργανώσεις, η ε, και οι κυβερνήσεις. Εμείς θα πρέπει ως Επιτροπή να το παρακολουθήσουμε πολύ στενά και τις εργασίες και τα αποτελέσματα αυτής της εταιρικής σχέσης. Και να έχουμε και μια επίσημη παρακολούθηση Ήδη, όπως γνωρίζετε, υπάρχουν, ε, υπάρχει μια ε, εταιρική σχέση της οποίας ηγείται η Σλοβακία ε, για τη στέγαση. Μια άλλη από την Ολλανδική, που, της οποίας ηγείται η Ολλανδική Προεδρία. Έχουμε τρεις τέτοιες εταιρικέ σχέσεις. από την αρχή, εξ αρχής όμως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να μην χάσει την ευκαιρία να παρακολουθήσει από πολύ κοντά την, ε, το έργο αυτών των εταιρικών σχέσεων, των συνεργασιών. Ε, ο ρόλος του Κοινοβουλίου βέβαια θα πρέπει να καθοριστεί σαφώς στο πλαίσιο του Συμφώνου του Άμστερνταμ. Δεν είναι σαφής ακόμα ο ρόλος των εκπροσώπων του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα διάφορα όργανα και τις δομές. Δύο ερωτήσει έχω να απευθύνω, όχι μόνο σε εσάς κυρία αλλά γενικότερα και στην Επιτροπή και μία παρατήρηση. Πρώτη ερώτηση. Πώς πιστεύετε, και ίσως αυτό είναι ένα ευχολόγιο, ε, σύμφωνα με το σύμφωνο του Άμστερνταμ και με το θεματολόγιο είναι σαφές ότι η διάσταση είναι οριζόντια, δεν αφορά τις περιφέρειες αλλά όλες τις, τις ε, περιοχές δράσης μας, καινοτομία, περιφερειακή πολιτική βέβαια, νέες τεχνολογίες, ε, είναι οριζόντια η θεματολογία αυτή. Πώς λοιπόν πιστεύετε ότι θα πρέπει να τη συντονίσουμε στην υλοποίησή της. Η, από την Επιτροπή είναι συναρμόδιοι τουλάχιστον πέντε επίτροποι. Οπότε τελικά στην πράξη ποιος θα συντονίζει την υλοποίηση η Κομισιόν είναι έτοιμη να ορίσει ένα συντονιστή, ένα μοναδικό συντονιστή. Ξέρω ότι είναι ρητορικό το ερώτημα, διότι όλοι γνωρίζουμε το πώς λειτουργούν τα πράγματα και τελικά κανείς δεν ξέρει ποιος θα το συντονίσει. Ποιος θα είναι συντονιστή στην πράξη. Και στο παρελθόν με το ψήφισμα μας ζητήσαμε συντονισμό και η απάντηση ήταν αόριστη. Παρ' όλα αυτά χρειάζεται κάποιος να το συντονίσει, κάποιος να συντονίσει την υλοποίηση. Δεύτερον, έχω τον εξή φόβο. Τι θα, δεν λέω θα τελειώσει η διαδικασία στο, το Μάιο, αλλά τι θα γίνει μετά τα τρία χρόνια. 2016 με 2018, ίσως και λίγο από το 19, Οπότε τα συμπεράσματα των εταιρικών σχέσεων θα είναι έτοιμα το 19 και τότε η πολιτική συνοχή θα πρέπει να είναι ήδη έτοιμη. Πώς θα ε, εξάγουμε συμπεράσματα και πότε θα εξάγουμε συμπεράσματα από τα τρία χρόνια έτσι ώστε να τα εντάξουμε στην πολιτική συνοχή, στη νέα πολιτική συνοχή. Οπότε μήπως θα πρέπει κατά τη διάρκεια των τριών αυτών ετών να προετοιμάζουμε εμεί σιγά σιγά την πολιτική συνοχής. Γιατί αλλιώς ε, προς τη μια μεριά θα κοιτάει η πολιτική συνοχής και προς άλλη μεριά τα συμπεράσματα των εταιρικών σχέσεων. Συνεπώς χρειάζεται ένα follow-up ε, των τριών ετών των συνεργατικών σχημάτων. Και μια παρατήρηση. Κάτι με το οποίο δεν συμφωνώ με τις ε, Eurocities με το δίκτυο. Ορισμένοι από μας ε, ε, εξακολουθούμε να διεκδικούμε μια πολιτική για τις πόλεις. Αυτό είναι ο ρόλος ο δικός μας ως πολιτικών. Θα πρέπει να, η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέτει μια πολιτική για τις πόλεις χωρίς να αντιβαίνει την αρχή της επικουρικότητας. Κάποιος θα πρέπει αργά ή γρήγορα να απαιτήσει ένα οριζόντιο εργαλείο που θα πρέπει να είναι η πολιτική για τις πόλεις, ανεξάρτητα αν τώρα μιλάμε για το θεματολόγιο μόνο. Ευχαριστώ. Thank you. Thank you very much, Mr. Van Ευχαριστώ, κύριε Βαν Νίστελρόι. Ναι. Αυτή η στιγμή είναι πολύ ωραία. Πριν από το σύμφωνο του Άμστερνταμ ε, κορυφώνεται το κύμα το οποίο σχηματιζόταν εδώ και δεκαετίες. Τώρα, το σύμφωνο μεταξύ άλλων μιλάει και για συμμετοχή. Έχουμε ένα πλαίσιο, αλλά εσείς θα πρέπει να δημιουργήσετε τη Συμμαχία των Προθήμων και να φροντίσετε για το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το σημαντικό στην ε, πολιτική. Δεν συμφωνώ απόλυτα με τον Γιάνν Όλμπριχ. Βεβαίω είναι μια ευρύτερη ατζέντα, αλλά στι συζητήσει μα για τη συνοχή στο μέλλον και την ενδιάμεση αξιολόγηση, γιατί να μην δούμε την ενσωματωμένη αυτή, την ολοκληρωμένη προσέγγιση όπως το κάναμε για τις περιφέρειες, την επικουρικότητα, τις συνθήκες. Και τώρα έχουμε κάποιες, κάποιους πυρήνες της πόλης στην Ευρώπη. Είναι πυρήνες τρόπων τεινά και μπορούμε να δούμε τι ισορροπία θέλουμε να υπάρχει μεταξύ των δύο επιπέδων. Η συζήτηση μπορεί να γίνει τώρα, δεν χρειάζεται να περιμένουμε τρία χρόνια. Υπάρχουν διάφορες πολιτικές στην Ευρώπη που επηρεάζουν το θεματολόγιο και η σημαντικότερη είναι η περιφερειακή ενδεχομένως που την συναποφασίζουμε εμείς. Είναι δικό μας θέμα. Χαίρομαι διότι έχουμε μια ισχυρή αντιπροσωπεία που θα πάει στο Άμστερνταμ για να γίνει συζήτηση με το Συμβούλιο γιατί αν στο σύμφωνο ε, είχα, είχαμε τη συνάντηση με την Επιτροπή των Περιφερειών, είχαμε συναντήσεις εδώ και τώρα είμαστε ένα βήμα πριν από το Άμστερνταμ. Και αν είμαστε ενωμένοι και εσείς θα είσαστε η εκπρόσωπός μας εκεί, και αν ε, δεν είναι η διατύπωση όπως πρέπει, εκεί πρέπει να μιλήσουμε. Η θέση του Κοινοβουλίου ε, δεν πρέπει να είναι ασαφής οι Ολλανδοί έχουν ήδη έναν εκπρόσωπο μέχρι τις 30 Μαΐου. Εμείς θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε μάχη για τη θέση μας και να συμβάλλουμε στην προετοιμασία, αν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Ε, πρέπει λοιπόν να ενισχυθούμε. Όχι ε, σε στιγμιαία μεμονωμένα θέματα, αλλά στα πλαίσια ενός γενικότερου σχεδιασμού πολιτικής. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Κοτσαλίνο. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε το Μάιο να τελειώσει η διαδικασία. Αντιθέτως, ξεκινάει μια καινούργια διαδικασία και πρέπει να ξεκινήσει μια πιο πλούσια, πιο δραστήρια περίοδος. Θέλω να κάνω και μια πρόταση προς, προς το δίκτυο τη, Ας αναζητήσει το δίκτυο τον τρόπο έτσι ώστε η αναθεώρηση και αξιολόγηση της πολιτικής συνοχής να συμπέσει με το θεματολόγιο έτσι ώστε να αλληλοσυμπληρωθούν και να λειτουργούν. Γιατί αλλιώς, ο διαχωρισμός μας φέρνει πάλι στο σημείο 0, στην αρχή. Έχουμε αυτά τα σχέδια δράσεων για τις πόλεις θα πρέπει να τα εγκρίνουμε αμέσω μετά το Άμστερνταμ. Και θα πρέπει να υπάρξει μια φάση ε, όπου ακούμε τις πόλεις. Να προσπαθήσουμε να αντιστρέψουμε λιγάκι τα πράγματα. Δηλαδή οι ίδιες οι πόλεις θα πρέπει να μιλήσουν. Θα πρέπει να υπάρξει ένας ε, συνασπισμός των πόλεων που θα μας βοηθήσει να σκεφτούμε μια νέα πολιτική συνοχής που θα ξεκινάει από κάτω και όχι από αποφάσεις που γεννώνται εδώ, από επιλογές που γίνονται εδώ, γιατί υπάρχουν διαγωνισμοί, γιατί υπάρχουν πολιτικές, υπάρχουν διευθύνσεις της Επιτροπής. Υπάρχει και μια κατεύθυνση σίγουρα. Ο Επίτροπος Πολιτικής Συνοχής, τουλάχιστον η άποψή μας είναι, θα πρέπει βεβαίως να παίξει ένα καθοδηγητικό ρόλο έτσι, ε, και να δώσει μια κατεύθυνση στην ε, πολιτική αυτή. Αλλά όμως και οι ίδιες οι πόλεις θα πρέπει να μιλήσουν. Ε, θα πρέπει δηλαδή μετά από 6, 7, 8 μήνε, ας πούμε, εμείς μαζί με την Επιτροπή, να δώσουμε ραντεβού με τι πόλεις για να δούμε πώ φαντάζονται το ρόλο του στη νέα πολιτική συνοχή μετά το 2020. Νομίζω ότι αυτό είναι ένας τρόπος για να δουλέψουμε μαζί σας και να μην ξοδέψουμε ας πούμε την ε, κληρονομιά που θα αφήσει το Άμστερνταμ. Είναι μια κληρονομιά που θα πρέπει να αξιοποιήσουμε, θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε από αυτής ε, τους επόμενους μήνες θα κλείσουν, μία, θα κλείσουν αυτόν τον κύκλο με συζήτηση και θα ανοίξει ένας νέος κύκλος όπου θα ακούμε περισσότερο τις α, αστικές περιοχές, τις ίδιες της πόλης. Θέλει κανένας άλλο τον λόγο. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τις ιδέες τους, για τις συνεισφορές τους, τη συζήτηση. Φυσικά είναι σημαντικό να βρούμε και το ρόλο που θα παίξει η δικιά μα η Επιτροπή, η Επιτροπή Ρέτζι και το ίδιο το Κοινοβούλιο στη διαδικασία αυτή. Διαδικασία που όλοι συμφωνούμε ότι δεν σταματάει στις 30 Μαΐου, αλλά συνεχίζεται. Και πρέπει να συνεχίσουμε μαζί με τα Εθνικά Κοινοβούλια, με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, μέσω των διαφόρων εκδηλώσεων, ε, ε, των διαφόρων ραντεβού ε, και με το EuroCities. Ελπίζω μέσα από αυτό το διάλογο να βρούμε τη σωστή κατεύθυνση. Στο εγγύς μέλλον θα έχουμε μία συνάντηση με τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων και θα μιλήσουμε για την αστική ατζέντα ε, και εκεί θα συνεχίσουμε τη συζήτηση και με τις Εθνικές Αρχές και με τους εκπροσώπους των πόλεων. Θέλετε να αντιδράσετε ή να πείτε κάποια καταληκτικά λόγια. Thank you. <clears throat> Just on... Ναι, ευχαριστώ. Για ένα-δύο σημεία. Για την πολιτική. Για τις αστικές περιοχές. Την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια τέτοια πολιτική. Πιστεύουμε σε αυτήν. Αλλά αν δεν υπάρχει σωστή διακυβέρνηση, δεν έχετε τα σωστά θεμέλια για να φτάσετε σε μια καλή πολιτική. Και αυτό λείπει, πιστεύουμε, αυτή τη στιγμή. Πέστε την governance, πέστε την πλαίσιο. Πρέπει όμως αυτό το πράγμα να το φτιάξουμε σωστά για να μπορέσουμε συνεχεία να πιέσουμε για να υπάρξει μια πραγματική πολιτική, για να υπάρξει αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα αστικά θέματα, για τα θέματα των πόλεων. Πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν, κατά την άποψή μου, ότι το πλαίσιο αυτό θα είναι πιο ισχυρό, ούτω ώστε να πείσουμε ότι έχουμε τα θεμέλια για να προχωρήσουμε. Για το ποιες πόλεις θα πρέπει να συμμετάσχουν, το είπαν κάποιοι συνάδελφοι. Το θέμα για μένα πάλι ανάγεται στη governance. Το θέμα δεν είναι να έχουμε 20.000 πόλεις, ούτε και ξέρω πόσες είναι στην Ευρώπη. Το θέμα είναι να υπάρχει διαφάνεια στις απόψεις και στις ιδέες, να υπάρχουν καλά κανάλια, ούτως ώστε να περνάνε τα μηνύματα από τις πόλεις, από την πραγματικότητα που ζουν οι πόλεις τέλος πάντων, μέσω αυτών των εταιρικών σχέσεων προς τα πάνω. Ούτως ώστε μέσα από τα το καναλιζάρισμα των μηνυμάτων, να δημιουργηθεί το απαραίτητο κονσένσου, η απαραίτητη συνένεση. Για μας το θέμα είναι να αξιοποιήσουμε αυτά που λέμε μέσα στο σωστό πλαίσιο. Δεν χρειάζεται να εφεύρουμε πράγματα γνωστά, να φτιάξουμε καλύτερα κανάλια επικοινωνίας, να είναι υποχρεωτικό η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη να περνάνε μέσα από αυτά τα κανάλια. Τα κανάλια αυτά, η διαφάνεια αυτή είναι απόλυτα απαραίτητη. Είναι πολύ σημαντικό, τουλάχιστον για τις 140 πόλεις, τις μεγαλύτερες πόλεις, αλλά είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τους υπόλοιπους εταίρους. Τρίτον, παρακολούθηση, η συνέχεια που δίδεται. Δεν είναι σημαντικό μόνο αυτά τα τρία χρόνια και ό,τι έχει γίνει, αλλά και το επέκεινα. Η πολιτική συνοχή είναι η πιο σημαντική πολιτική που η μέθοδος της, ε, του αστικού θεματολογίου μπορεί να εφαρμοστεί. Δηλαδή να γίνει σεβαστή η αστική διάσταση στην πολιτική συνοχή. Αλλά υπάρχουν και όλοι οι άλλοι τομεί, όπω είπατε. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι σε ό,τι αφορά την νομοθεσία και τη χρηματοδότηση, έχουμε τώρα την ενδιάμεση αναθεώρηση του προπολογισμού. Να εξασφαλίσουμε λοιπόν ότι τα αποτελέσματα και τα μηνύματα των, που θέλουν να διαμηνήσουν οι πόλεις φτάνουν ως τις τομιακές πολιτικές και απεικονίζονται σε αυτό. Και με αυτόν τον τρόπο και οι υπόλοιπε κοινοβουλευτικέ επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, μπλέκονται περισσότερο. Και η ομάδα μας παίζει το μεγαλύτερο λόγο. Ας πούμε για την ποιότητα του αέρα, ε, εκεί παίζει το ρόλο της η Επιτροπή ΕΜΒΗ. Θα πρέπει να υπάρχει αυτή η οριζόντια διάσταση, τα σωστά άτομα να εμπλέκονται τα σωστά υπουργεία, όχι μόνο τα υπουργεία ας πούμε, αστικού σχεδιασμού, αλλά όλα τα άλλα υπουργεία, ας πούμε, για την Επιτροπή Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Περιβάλλοντος κτλ. κτλ. Για μένα όλα αυτά είναι πολύ σημαντικό. Η σχέση με τη συνοχή, για να πάω σε αυτό το κομμάτι, και εκεί έχω να στείλω κάποια μηνύματα. Η συνοχή έχει το δεύτερο μεγαλύτερο προϋπολογισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν πάρα πολλές επενδύσεις που αφορούν τις πόλεις εκεί, από την πολιτική συνοχή. Και υπάρχει μια βελτίωση από περίοδο προγραμματισμού σε περίοδο προγραμματισμού. Χάρη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που πίεσε, ε, τα μέλη της Επιτροπής σας αλλά και άλλους πιέσατε ούτω ώστε να έχουμε μια ισχυρότερη αστική διάσταση στην πολιτική συνοχή. Αλλά δεν είμαστε στο ιδανικό επίπεδο ακόμα. Καταρχάς πρέπει να δούμε πού πάει η πολιτική συνοχή. Και το πρώτο μήνυμά μου είναι ότι πρέπει να έχουμε το σωστό χρονισμό. Δεν θέλω να πω ότι χάσαμε το τρένο, ότι είναι πολύ αργά. Είναι πολύ περίεργο γιατί αυτή τη στιγμή, δύο χρόνια μετά την έγκριση του καονισμού, αρχίζουν οι, ε, οι να ξοδεύουν λεφτά. Το βλέπουμε κάθε μέρα στι περιφέρειε στι πόλει κτλ. Αν δεν τα κάνετε σωστά τώρα, να σκεφ... αν δεν σκεφτείτε τώρα την πολιτική, την δομή, του κανονισμού που θέλετε, θα καταλήξετε να, ζει... να ζείτε ξανά αυτά που ζούμε τώρα. Δηλαδή, μια καταστροφή σε σχέση με την εφαρμογή. Έχουμε απίστευτε καθυστερήσει. Καθυστερεί ο δεύτερο κανονισμό. Ο κανονισμό για τι ε, εκτελεστικέ και εφαρμοστικέ πράξει δεν είναι έτοιμος. Επομένως, ε, όλα τα εργαλεία του δημοσιονομικού μηχανισμού δεν υπάρχουν. Κανονικά όλα θα έπρεπε να είναι τώρα στο τραπέζι. Ήδη εφαρμόζεται την αστική, το αστικό θεματολόγιο στην πολιτική συνοχής. Μας ακούτε δηλαδή εμάς. Σωστό είναι αυτό, αλλά πρέπει να καταλάβετε και τι θέλουμε. Επομένως, το πρώτο μου μήνυμα είναι αν θέλετε μια τελείως διαφορετική πολιτική συνοχής, προσοχή, προσοχή. Προσοχή την εφαρμογή της. Εγώ ζω την πραγματικότητα αυτών που καλούνται να εφαρμόσουν τις πολιτικές και πραγματικά ο βίος τους γίνεται δύσκολος. Είναι ασύλληπτα δύσκολο το να δημιουργήσουμε τα συστήματα το σύστημα ελέγχων, το σύστημα διαχείρισης. Τα τελευταία δύο χρόνια πέρασαμε με έναν εφιάλτη. Αν έρθετε εδώ και μας πείτε ότι η πολιτική συνοχή θα αλλάξει άρδιν, θα γίνει επανάσταση. Κανένα δεν θέλει να ξοδεύει λεφτά από την πολιτική συνοχή πια. Είναι ασύλληπτα δύσκολο να βρούμε δικαιούχου που να θέλουν και να μπορούν να ξοδέψουν τα λεφτά τη πολιτική συνοχή. Πρέπει να εξασφαλίσουμε μια σωστή αλλαγή. Η αλλαγή θα είναι 100% εκθεμελίων ας πούμε, εξαφανίσετε την πολιτική συνοχής ή θα πρέπει να αλλάξετε τις προτεραιότητες, θα κάνετε πιο ευέλικτα πράγματα, γιατί τώρα εξετάζουμε τι γίνεται με την προσφυγική κρίση και πώς μπορούμε να προσαρμοστούμε και δημιουργεί, μας δημιουργεί ασύλληπτες δυσκολίες. Όλη αυτή η μεικτή διαχείριση δημιουργεί ατελείωτες δυσκολίες. Είναι ένα άλλο μήνυμα. Not... Ας επωφεληθούμε από αυτά που έχουμε, ας τα αξιοποιήσουμε πριν τα πετάξουμε στον κάλαθο των αχρήστων. Η Κομισιόν ψάχνει και άλλους τρόπους για να χρησιμοποιήσει την πολιτική συνοχής. Κυκλοφορούν έτσι ανεπίσημα διάφορες ιδέες να δώσουν τη χρηματοδότηση, τα ποσά δηλαδή στα κράτη-μέλη, ούτω ώστε να φτιάξουν τι δικέ του ε, μεταρρυθμίσει και τη δική του μεταρρυθμιστική πολιτική. Δεν ξέρω τι άποψη έχετε γι' αυτό. Πρέπει να αρχίσετε όμως, πρέπει να αρχίσετε κι εσείς να παίζετε κάποιο ρόλο πιο έντονο ας πούμε για την πολιτική συνοχή. Τώρα για το αστικό κομμάτι θα σας πούμε κάτι πολύ προφανές. Για μας η πολιτική συνοχής πρέπει να γίνει πιο αστική εντό αγωγικών. Ε, ήταν, ένα, ήταν αστική κάτω το 20%. ελάχιστο 5, το πολύ 20, αλλά εμείς θέλουμε περισσότερο από 20%. Και περισσότερη χώριση στις πόλεις, στους φορείς των πόλεων, πειράματα, όπως το ITI, η απευθείας εκχώρηση αρμοδιοτήτων είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο αν θέλουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Γιατί αυτό δεν συμβαίνει σήμερα, δεν υπάρχει, μας λείπει. Ξοδεύουμε για το αστικό κομμάτι, αλλά δεν υπάρχει καμία ολοκλήρωση, ας πούμε. Εταιρική σχέση, άλλο στοιχείο. Αν θέλετε να παίξετε σωστά το ρόλο σας, και δεν θα σας πω ότι ξανά ότι το 75% του πληθυσμού ζει στις πόλεις, γιατί είναι βαρετό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν θέλετε ανταγωνιστική Ευρώπη, οι πόλεις παίζουν σημαντικό ρόλο. Εάν θέλουμε να έχουμε μια πολιτική συνοχή που είναι πιο αστική, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να φτιάξουν τις ε, συμφωνίες εταιρικής σχέσης και τα επιχειρησιακά προγράμματα πιο ευθυγραμμισμένα με τις ανάγκες των πόλεων. Σήμερα έχουμε επιλογή των έργων, έχουμε τον κώδικα διοντολογίας που έγινε στα τα κρατήματα μπορούν να αποφασίσουν αν θα έχουν ITIs ή όχι. Χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω. Σχεδόν τελείωσα. Καινοτόμε δράσει. Ε, είδατε πόσε πόλει ε, ανταποκρίθηκαν σε αυτή την έκκληση. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνει η καινοτομία στις πόλεις ή θα καινοτομήσουν οι πόλεις. Χωρίς ε, τα επαχθή ε, εργαλεία και μηχανισμούς της χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Yeah, Ολοκληρωμένη προσέγγιση, εταιρική σχέση και, και, και... Νομίζω τα είπα, τα βασικά. We are totally available and Είμαστε στη διάθεσή σας πάντως, ανοιχτή, διαθέσιμη για ανταλλαγές σε κάθε επίπεδο. Και τεχνικός πώς και αλέος πώς για να σας ε, μιλήσουμε για τις εμπειρίες μας από την εφαρμογή των διαρθωτικών ταμείων, τι δουλεύει, τι δεν δουλεύει με αυτά, το βασικό είναι ότι χρειαζόμαστε μια πολιτική συνοχής ανοιχτή για όλα τα εδάφη, όλους τους χώρους, πόλεις και μη, αλλά περισσότερη αστική διάσταση. Και η αστική διάσταση να συνδέεται με, τον, με την ύπεθρο. Θέλουμε καλύτερη σχέση δηλαδή αστικού, και, αστικού χώρου και υπαίθρου. Αυτή η σύγκρουση δεν είναι για κανέναν ολοκληρωμένη διαχείριση και διαχείριση απευθείας από πόλεις οι αστικές περιοχές, με πραγματικές εταιρικέ σχέσεις, με καλύτερη συνεργασία και με τις περιφέρειες για την ανάπτυξη των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Και τελευταίο και σημαντικό, όλα να γίνουν απλούστερα. Είμαι μέλος της ομάδας για την απλούστευση των διαφορετικών ταμείων για τους ε, δικαιούχους και σας λέω ότι υπάρχουν τρει-τέσσερι τομεί άκρο πολιτική που πρέπει να του ξαναδούμε. Το θέμα των ελέγχων, κρατικέ ενισχύσει, το θέμα του χρονισμού, ο πρωτογενή νομοθεσία και η δεύτερογενή νομοθεσία. Μπορώ να μιλάω ολόκληρη τη μέρα, αλλά δεν είμαι εδώ γι' αυτό. Είμαι στη διάθεσή σας, όποτε το επιθυμείτε, να κάνουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων και βασίστετε πάνω μας θα σας δώσουμε την άποψη των πόλεων. Thank you. Thank you very much. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σήμερα ως ε, τμήμα της ε, ε, διαδικασίας εξακρίβωσης αλλά και της προετοιμασίας μας για την έναρξη της συζήτησης για την μελλοντική πολιτική συνοχής. Χτες συζητήσαμε αρχικά το μέλλον του πολιτισμού δημοσιονομικού πλαισίου, την αναθεώρησή του κλπ. Ακούσαμε σήμερα εσάς, σκεφτόμαστε να τοποθετήσουμε το θεματολόγιο για τις πόλεις ε, στο επίκεντρο της μελλοντικής πολιτικής συνοχής. Βρισκόμαστε στο, το μέσο της συζήτησης αυτής, οπότε ε, βρίσκεστε στο σωστό χώρο τη σωστή στιγμή. Ελπίζω ότι θα εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας και ελπίζω ότι θα συμμετάσχετε και σε μελλοντικέ μας συνεδριάσεις με διάφορες μορφές έτσι ώστε να συζητήσουμε την μελλοντική πολιτική συνοχής και το ρόλο των πόλεων σε αυτήν. Αν δεν έχετε άλλες προτάσεις, ε, αν δεν έχετε, αν υπάρχει κανείς άλλος που να θέλει το λόγο να ρωτήσει την κυρία Μπόνη οτιδήποτε, σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε κυρία Μπόνη. Συνεχίζουμε. Το επόμενο σημείο είναι η έγκριση των προαποφάσεων των συντονιστών. Οι συντονιστές συνήλθαν χτες και οι αποφάσεις τους σας εστάλησαν με email. Τις εγκρίνετε. Ωραία. Ναι. Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Διάφορα. Υπάρχει κάτι στα διάφορα. Όχι. Ωραία. Οπότε να επωφεληθώ για να σας υπενθυμίσω πως έχει προγραμματιστεί μια συνάντηση για, το, για το ρόλο των περιφερειών στην λήψη των αποφάσεων οργανώνεται από το ΕΛΚ σήμερα στις 5.30 το απόγευμα θα λάβει χώρα στο, στην αίθουσα ανάγνωσης της ε, βιβλιοθήκης ο κ. Βάλτεστελ θα κάνει τις αρχικές ε, εισαγωγικές παρατηρήσεις και θα έχουμε και διάφορους ομιλητές μεταξύ αυτών την κυρία Χούμπνερ. Αυτά για σήμερα. Σας υπενθυμίζω ότι η επόμενη συνεδρίαση είναι, θα λάβει χώρα την 3η 24 Μαΐου το απόγευμα. Μισή μέρα λοιπόν Ευχαριστώ πολύ τους διερμηνείς, λέει πρόεδρος. Ευχαριστώ όλους και όλες. Λήξη της συνεδρίασης.